Καλημέρα σας. Ήρθατε ακριβείς όλοι. Ωραία. Χθες το βράδυ μας δυσκόλεψε η συνάντηση των συντονιστών. Δεν έφταιγαν εκείνοι, αλλά τα θέματα. Από το ίντερνετ ίσως χθες το βράδυ μάθατε τα αποτελέσματα. Πρόκειται για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας και θα δούμε εκεί τι θα γίνει τελικά, γιατί η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ζήτησε έκθεση πρωτοβουλίας στην συνεδρίαση των Πρόεδρων Επιτροπών για τον πλουραλισμό των μέσων και χθε το βράδυ ε, είπαμε ότι αυτό δεν είναι θέμα Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, είναι κατεξοχήν θέμα δικό μας. Είμαστε υπεύθυνοι για τα οπτικοακουστικά, για τα ΜΜΕ, υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Τι συμβαίνει, δεν έχετε διερμηνία. Εκεί εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Και με τους ε, συντονιστές, με μία εξαίρεση, όλοι οι άλλοι συμφώνησαν ότι θέλουμε εμείς να το αναλάβουμε. Αν κερδίσουμε τη μάχη αυτή, και εγώ θα κάνω το παν για να κερδίσουμε, τότε θα πρέπει ε, εδώ να γίνει η έκθεση. Η έκθεση πρωτοβουλίας που συμφωνήσαμε χτες, οι εκθέσεις θα πρέπει να αναβληθούν, μία τουλάχιστον. Ενημερωτικά. Έχουμε μάχη, η Λίμπε θέλει μόνη της, άρχισε από το νομοσχέδιο της Ουγγαρίας για τα ΜΜΕ. Εμείς πρέπει να προσέξουμε, να μην μας παίρνουν τη δουλειά τη δική μας οι άλλοι. Αν θέλουν να γνωμοδοτήσουν, παρακαλώ για το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εκείνοι αναφέρονται στο άρθρο 162 νομίζω του χάρτη και ότι λένε ότι είναι υπεύθυνοι να φροντίζουν για τα πρότυπα που θα διέπουν την ελευθεροτυπία του τύπου. Αν έχει να κάνει με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι και δική μας δουλειά και της ΛΥΜΠΕ. Γιατί η ΛΥΜΠΕ ένα κομμάτι μόνο ε, παρακολουθεί. Ενώ εμείς είμαστε εξοχήν υπεύθυνοι. Σας υπόσχομαι λοιπόν ότι θα τσακωθώ για αυτό το θέμα. Και αν κερδίσω το, τη διαμάχη αυτή, που το υποθέτω, θα καταπιαστούμε με αυτή την έκθεση πρώτα και η Μπολόνια, που είπαμε ότι θα το κάνουμε χθε, θα ακολουθήσει. Όλα τα άλλα θα τα διαβάσετε στα πρακτικά που νομίζω χθε το βράδυ εστάλησαν. Για τις ψηφοφορίες Τώρα, Youth on the Move, έχουμε να το ψηφίσουμε. Υπάρχουν προβλήματα, μιλάν, όλα εντάξει, όλα εντάξει. Πάμε στην ψηφοφορία. Πάρτε την κάρτα σας, έχετε την έτοιμη γιατί μπορεί να έχουμε δυσκολίες. ΕΛΚ 14. 2, δεν πρέπει να... Ποιοι θα... Ήβο και Μάτουλα. Εντάξει. Αποσύρονται εθελοντικά. Ευχαριστώ. Θα προσέχουμε. Πάντως έχουν μεγάλη επιτυχία στην προσέλευση. Είναι πάντα εδώ. Πρωτοπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ Α, 13 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας 9 υπέρ 13 κατά απορρίπτεται η 15 ήταν αυτή. 16. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18. Υπέρ όχι, 19 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 20 υπέρ, κατά, αποχές, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τώρα πέρας. Απορρίφθηκε 10 προς 16. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 και 115 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτές 28 και 29 υπέρ κατά αποχές δεκτές προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 32 σε δύο μέρη πρώτο τμήμα της 32 κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 προς 13 απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 35. Μόνο για τα αγγλικά. 36 υπέρ. Κατά. 36 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 37 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12 προς 14 απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται. Τις 42 πέρα στις ψηφοφορίες. 12 προς 13 απορρίπτεται 46, 48 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές δεκτές 47 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 9. Έμπλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 20. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε αυτό άρχεται η ψηφοφορία πέρας 12 προς 12 απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 αποσύρθηκε 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 68-69 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτές πέντε προφορική τροπολογία πέντε υπέρ κατά αποχές δεκτή Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα αν εγκριθεί. Πάμε στην, προφορική έξι. 6 λοιπόν προφορική υπέρ κατά δεκτή. 74. Α, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε αυτό άρχεται η ψηφοφορία για την 75 πέρας 17 προς 11 δεκτή. «76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται». «78 υπέρ κατά αποχές δεκτή». «77 υπέρ». Α, όχι, απορρίφθηκε 78, υπερ κατα αποχες δεκτεί. 77 οχι κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 της έμπουλ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 προς 14 απορρίπτεται. Έμπλ 2. Υπέρ. Κατά. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε 14 προς 14. 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 86 υπέρ κατά έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. 86 ψηφίζεται. Πέρασε. 11 προς 16. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία. Εγώ ήθελα να πω ότι είμαστε κατά. Θα ενημερώσετε την ομάδα, το πείτε στην ομάδα. Ο προφορική 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 90 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 92 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 της έμπλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 100 υπέρ κατά ξανά υπέρ ευχαριστώ κατά αποχές δεκτή 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή καλή γυμναστική άμα το κάνετε και λίγο πιο έτσι με ζέση είναι καλό για το σώμα 103 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 106 υπέρ κατά αποχές δε ξανά υπέρ Ωραία, με χρονοκαθυστέρηση λειτουργείται καμιά φορά. 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 109 υπέρ κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκαεφτά προς 10 δεκτή. Αυτή ήταν η 109. Πάμε τώρα στην 110, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 111, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 της έμπουλ υπέρ κατά ξανά 10 ψηφίζουμε τη έμπουλ υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 έμπουλ υπέρ κατά αποχές δεκτή 123-134 υπέρ κατά αποχές δεκτές 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας 14 προς 14 απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή 137, 141 υπέρ κατά αποχές δεκτές 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτό να το ελέγξουμε. Το δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 10 προς 19 απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται πέρας 19 προς 8 δεκτή Εκατόν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 146 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 153 υπέρ κατά κανείς δεκτή λοιπόν, 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 155 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές δεκτή 160 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας 20 προς 8. Καλή γυμναστική. 161 Μάρκο υπέρ κατά αποχές δεκτή. 162 υπέρ. Είναι για διαγραφή. Αν θα διαγραφεί ή όχι. Είναι για το περιεχόμενο αφορά. Είναι το περιεχόμενο. Προσέξτε. 162 υπέρ. Κατά. Θαυμάσια απορρίφθηκε. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 29 έμπουλ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ΕΜΠΛΕΝΑ, υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 προς 13 δεκτή. 168. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 170 σε τέσσερα τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τέταρτο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 προς 14 δεκτό. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 172, 175 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 173 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλ 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή έμπλ 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή 179 υπέρ κατά αποχές δεκτή, έμπλ 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 180 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 181 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 182 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 183-184 έχουν καλυφθεί από το έμπλεμα. 185 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 189 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 19 της έμπλ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 192 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 α όχι αποσυρθεί και 198 υπέρ κατά αποχές δεκτή 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 202 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 205 καλύφθηκε ήδη από την έμπλ 16 206 υπέρ κατά αποχές δεκτή 207 υπέρ κατά αποχές δεκτή 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 211 υπέρ, κατά έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 11 προς 14. 212. Όχι. Δο, ναι. 212 υπέρ. Κατά αποχές άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρας. 15 προς 14. Δεκτή. 213. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 218. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απεσύρθη 215-216 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 217 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 219 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 223 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 224 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές δεκτή 220 απεσύρθη 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Μάλιστα. τελική ψηφοφορία δεν χρειάζεται όχι πώς άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. «27 υπέρ, μόνο δύο αποχές, ε, θερμά συγχαρητήρια Μίλαν Σβέρ». Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες για την ψηφοφορία. Θα ήθελα επίση να σα ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας στη σύνταξη του κειμένου και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο και την Πέτρα που με βοήθησαν στο φάκελο αυτό. Ευχαριστώ Μίλαν. Πάμε στο σημείο 10 της ημερήσια διάταξης πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριος Ιβαν δεν είναι εδώ. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να πει τίποτα. Περνάμε άμεσα στην ψηφοφορία. Καφέ.

Αρχίζουμε λοιπόν με την τροπολογία 1 υπέρ κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. 17 προς 9. Λοιπόν, στα γρήγορα να τελειώνουμε. 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ α καταπίπτει 11 λοιπόν υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό ή 13 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας 12 προς 17 απορρίπτεται η 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 36 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Συμβιβαστική. Στην παράγραφο 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές δεκτό 53 υπέρ αποσύρθηκε αλλά δεν το λέει ο κατάλογος 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία επί της 51 πέρας 16 προς 13 δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά θα το κάνουμε υπέρ άρχεται ψηφοφορία όχι άρχεται ψηφοφορία απλώς πέρας 27 προς 2 Αποχές δεν έχει. Συγχαίρουμε τον Απόντα Ιβάν. Σημείο 11. Συνολική προσέγγιση. Κύριε Κέλλη, θέλετε να πείτε στην αρχή τίποτε. Τίποτε. Αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία στην 6. Πέρας. 10 προς 19 απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ Μπεναράμπα του προφορική. Έπρεπε να είχατε σηκώσει το χέρι. Ναι, θα μιλήσω τονίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στον εργοδότη και αφορά την επαγγελματική κατάσταση των χρηστών δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται ή να προωθούνται σε κάποιο τρίτο μέρο χωρί την προηγούμενη ε, ε, άδεια του... χωρίς την προηγούμενη άδεια του ε, αναφερόμενου ατόμου. Τα στοιχεία τα προσωπικά του, τα οποία προωθούνται στον εργοδότη του, δεν θα πρέπει να προωθούν σε τρίτο άτομο χωρίς προηγούμενη συνένεση του ενδιαφερόμενου. Το υπαρθμόν 11 δεν είναι το σύνολο της τροπολογίας, είναι μια προφορική τροπολογία στην τροπολογία υπαριθμών 11. Σωστά? Ναι, στην 11 ακριβώς. Λοιπόν, θέλετε... Τι θέλετε ακριβώς? Θέλετε να προσθέσετε λοιπόν ναι, που του στον εργοδότη. Ναι, ακριβώ. Διάβασα την τελική εκδοχή αυτού του τμήματο, συμπεριλαμβάνοντα και την φράση αυτή. Εκτό μικροφώνου, πρόεδρο. Εκτό μικροφώνου, πρόεδρο. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 11 με την προσθήκη αυτή που επικοινωνείται στον εργοδότη. Να το διαβάσετε άλλη μια φορά. Η τροπολογία είναι η ακόλουθη, τελική εκδοχή της. Τονίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία τα οποία επικοινωνούνται στον εργοδότη και που αφορούν στην επαγγελματική κατάσταση του χρήστη δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται ή να προωθούνται σε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη άδεια του ενδιαφερόμενου ατόμου, του εν λόγω ατόμου. Ναι, είναι αποδεκτό. Είναι αποδεκτή. Καλώς. Τροπολογία 11 λοιπόν, με την καινούργια μορφή υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή. Είχατε τύχη που τα αλλάξατε, γιατί πριν ήταν κατά. 12 υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται, η 15 αποσύρθηκε, 16 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 18 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 21 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 δύο μέρη πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Προφορική της Νάντια Χίρς. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 34 υπέρ κατά αποχές δεκτό τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας 29 προς 0 καταπληκτικό όλα τα μέτρα της Ιρλανδικής κυβέρνησης την ίδια τύχη να έχουν. Θέλετε να πείτε κάτι. Να ευχαριστήσω όλους μόνο για την υποστήριξη. Ευχαριστώ και σας κυρία Πρόεδρε γιατί σήμερα ε, υιοθετήσατε πολύ αποτελεσματικό σύστημα στις ψηφοφορίες. Πάμε στο σημείο 12 που δεν υφίσταται όμως γιατί η κυρία Βασιλείου δεν είναι εδώ διότι ε, κάποιος από την οικογένεια ε, πέθανε, δεν μπόρεσε να έρθει. Πάμε στο σημείο 13 λοιπόν της ημερήσιας διάταξης έκθεση. Ή, ήσυχα εκεί οι συνεργάτες. Κάνει τρομερή φασαρία. Κύριε Παπα-Νικολάου. Η ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού. Ξέρετε ότι επιτέλους κερδίσαμε αυτό που ζητούσαμε από την έκθεσή μου το 96 υπάρχει στη συνθήκη ο αθλητισμός αλλά θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε αυτό και υπάρχει μια ανακοίνωση της Κομισιόν και ο συνάδελφος ε, Σαντιάγκο Φίσας ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Γι' αυτό θα του δώσουμε το λόγο για να μας πει τις πρώτες εντυπώσεις του, τι θα κάνει. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την Επίτροπο Βασιλείου για την εξαιρετική εργασία που έχει φέρει σε πέρας ως προς την ανακοίνωση της περασμένης Πέμπτης για την Ευρωπαϊκή Διάσταση του Αθλητισμού. Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί την Λευκή Βίβλο του 2007 και σέβεται και τις νέες δικαιοδοσίες που δίνει το άρθρο 155 της Συνθήκης της Λισαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω την τιμή να είμαι ο εισηγητής με στόχο της έκθεσης να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε λίγο παραπάνω σε αυτή την προώθηση της Ευρωπαϊκής Διάστασης Δελτισμού και να δημιουργηθεί ένας διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και άλλες επιτροπές που ενδιαφέρονται για την έκθεση αυτή και ότι έχουμε επομένως κοινά συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Η Επιτροπή μας καθώς και το ΕΛΚ έχουν, είχαν οργανώσει μία ακρόαση τον Μάρτιο από την οποία εποφεληθήκαμε και ευχαριστώ τους σοσιαλιστές συναδέλφους που συμμετέσχουν στην ε, ακρόαση αυτή που οργάνωσε η ομάδα μου. Λοιπόν, πρώτο θέμα που τίθεται είναι η επικουρικότητα. Το αναφέρει η ανακοίνωση ρητά αναγνωρίζεται δηλαδή η δικαιοδοσία των χωρών μελών για τον αθλητισμό. Θα ήθελα όμως επίσης να τονίσω την ιδιαιτερότητα που έχει ο αθλητισμός και που την αναφέρει το άρθρο 165. Η Κομισιόν δεν αγνόησε τις ιδιαιτερότητες αυτές του αθλητισμού επιμένοντας ιδιαίτερα στην κοινωνική του και εκπαιδευτική του διάσταση καθώς και στον εθελοντικό του χαρακτήρα. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά περιγράφουν τον αθλητισμό. Οι αθλητικές οργανώσεις χρειάζονται τη βοήθεια της Ένωσης για να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως το ντοπάρισμα και για να διατηρήσουν τη δομή των αθλητικών δραστηριοτήτων η Λευκή Βίβλος επιβεβαίωσε ότι η ενωσιακή δράση στον τομέα αυτών μπορεί να προσφέρει πολλά. Και στην ανακοίνωσή της αν χωρίζεται σε τρία τμήματα, στην δε έκθεσή μου τα επαναλαμβάνω κι εγώ, προσθέτοντας όμως και το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Πρώτο τμήμα, ο κοινωνικός ρόλος του αθλητισμού, δηλαδή το νόημα που έχει για την κοινωνία. Δεύτερον, η οικονομική του διάσταση, δηλαδή η συνεισφορά του αθλητισμού στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Τρίτον, η οργάνωση του και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί αθλητικοί παράγοντες έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν στην οργάνωση του αθλητισμού. Θα ήθελα να επιμείνω ιδιαίτερα στον κοινωνικό ρόλο όμως. Καταρχήν ότι είναι εθελοντικός ο χαρακτήρας του. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό στον αθλητισμό. Χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν εθελοντικά στον αθλητισμό, πράγμα που επιτρέπει τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων στην Ευρώπη. Ο εθελοντικός χαρακτήρας είναι ανοιχτό σε όλους, σε όλες τις ηλικίε φύλλα και εθνότητες ή προέλευση. Θα θέλαμε λοιπόν να πατήσουμε φόρο τιμή σε όλους όσους και όλες όσες συνεισφέρουν στον αθλητισμό εθελοντικά. Η καταπολέμηση του τοπαρίσματος είναι μεγάλη πρόκληση για όλους τους αθλητικούς παράγοντες. Οι τοξικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι μεγάλη πληγή του αθλητισμού και αφορά και τον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό. αντιμετωπίζουν μεγάλους κινδύνους όσοι το πάρονται. Υπάρχει ολόκληρο δίκτυο οργανωμένο και η έλλειψη πληροφόρησης για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ντοπαριζόμενοι είναι κάτι ακόμα πιο επικίνδυνο. Το άρθρο 83.1 της Συνθήκης Λισαβόνας μας επιτρέπει να διώξουμε διοσκαστικώς τους υπευθύνου. και χωρίς να παραγνωρίσουμε καθόλου το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των αθλουμένων. Θα ήθελα να επιμείνω στον θετικό χαρακτήρα που παίζει ο αθλητισμός στα σχολεία, διότι διευκολύνει την αλληλεγγύη και τη φιλία μεταξύ προσώπων από διαφορετικές κατηγορίες και ομάδες. Πρέπει λοιπόν από την αρχή να επιμένουν τα σχολεία στον αθλητισμό διότι έτσι θα αποφευχθούν πληγές όπως ε, η τοξικομανία και ο αλκοολισμός. Άλλο θέμα η παιδεία. Έχουμε δει από την ακρόαση ότι μπορεί να, υπάρχουν, να υπάρχει διπλή καριέρα των αθλητών σε πολλές χώρες και αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη λήψη διάφορων μέτρων. Είναι ουσιώδες κατά την αθλητική του σταδιοδρομία να μπορεί κανείς να παρακολουθεί ταυτόχρονα μία ποιοτική εκπαίδευση για να έχει κάποτε μία μόνιμη θέση στην αγορά εργασίας. Πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν τις σπουδές τους οι αθλούμενοι χωρίς να παραγνωρίζει μία σταδιοδρομία την άλλη. Γι' αυτό πολλά πανεπιστήμια έχουν προβλέψει και ειδικά προγράμματα για όσους θέλουν να ασχοληθούν ιδιαίτερα με τον αθλητισμό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες για να προσαρμόσουμε τα προγράμματα, παραδείγματος χάρη της Βολονίας, σε περισσότερο αθλητισμό να προταθούν ε, εκπαιδευτικά προγράμματα και μέσω του ίντερνετ. Τώρα, η βία στον αθλητισμό, δυστυχώς ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και η ομοφοβία υπάρχουν και στον αθλητισμό. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ενδυναμώσουμε τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και να αναλάβουμε και νέα για να καταργήσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πληγές του αθλητισμού. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερα και γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερος. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τα ωφέλη που αποφέρει ο αθλητισμός για τη δημόσια υγεία. Είναι βασικό αγαθό, μπορεί να αποφύγει τις παιδικές ασθένειες που οφείλονται στην καθιστική ζωή. Ο αθλητισμός σημαίνει ευημερία και υγεία και διαπιστώνουμε ότι η άθληση ωφελεί όχι μόνο τον ενεργό πληθυσμό αλλά και τους συνταξιούχους. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να ασχολούνται με σωματικά και πνευματικά σπορ έτσι ώστε άρα μάλλον χρειάζεται προώθηση του αθλητισμού και στους ηλικιωμένους. Θα ήθελα επίσης να επιμείνω σε άλλα ωφέλη του αθλητισμού. Μπορεί να αποτελέσει στοιχείο συμπερίληψης και ολοκλήρωσης μειονοτικών ομάδων ή περιθωριακών ομάδων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη γυναικεία του διάσταση τόσο ως προς την άθληση όσο και προς την εξάσκηση των αθλουμένων την γύμναση. Πρέπει να προωθήσουμε το γυναικείο αθλητισμό λοιπόν. Με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω την προώθηση από τις αθλητικές ομοσπονδίες των δραστηριοτήτων για τους αναπήρους και επίσης την υποστήριξη και προώθηση των ειδικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν αυτοί. Ο αθλητισμός παίζει ένα σημαντικό οικονομικό ρόλο, αλλά οι περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες δομούνται πάνω στον εθελοντικό τους χαρακτήρα και τίθεται επομένως το θέμα της χρηματοδότησης. Πρέπει να δοθεί χρηματοδότηση και κεντρικά στον αθλητισμό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας ή διανοητικής ιδιοκτησίας στον αθλητισμό, ώστε να μπορεί ο αθλητής να έχει κάποια αποζημίωση αν δεν γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα που αφορούν να μεταδώσεις, παραδείγματος χάρη. Αν οι οργανωτές μπορούν να επιλέγουν ποια επιχείρηση θα αναμεταδώσουν, θα μπορούσαν να αποφευχθούν πολλά προβλήματα. Έπειτα για τα δικαιώματα αυτά αναμετάδοση συγκεκριμένα πρέπει να υπάρξει μία αρχή αλληλεγγύη και σε αυτό υπέρ του αθλητισμού. Δηλαδή ιδιαίτερα να επιμείνουμε στη θετική επίπτωση που έχει ο αθλητισμός στην οικονομία και μάλιστα σε πολλούς οικονομικούς τομείς. Η υποστήριξη του αθλητισμού πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα διαρθρωτικά ταμεία. Και τώρα, το τέταρτο κεφάλαιο για την ανάπτυξη του αθλητισμού τίθεται το θέμα της καλής διακυβέρνησης και στον αθλητισμό γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αυτονομία και την καλή διαχείριση των αθλητικών οργανώσεων. Η αυτονομία, η δημοκρατία, η διαφάνεια, η ευθύνη, η υπευθυνότητα και μία σωστή και ισορροπημένη εκπροσώπηση είναι οι αρχές που διέπουν την καλή διακυβέρνηση. Έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα για τέτοια καλή αθλητική διακυβέρνηση και έτσι θα μπορούσαμε με τη γενίκευσή τους να ωφελήσουμε τον αθλητισμό γενικότερα. Υπάρχει και το θέμα της ελεύθερης κυκαλοφορίας. Έχει βέβαια τις ιδιαιτερότητες του αθλητισμού, Πρέπει να στηρίξουμε τις εθνικές δομές και τις εθνικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται πανενωσιακώς. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει κάποιος έλεγχος των μεταγραφών έτσι ώστε να μην σπαταλούνται τα χρήματα που διατίθενται για αυτόν. Το σύστημα της FIFA που λέγεται TMS είναι σύστημα βάση του οποίου οι αθλητικοί σύλλογοι υποχρεώνονται να πληρούν περίπου 30 κριτήρια για να εγκριθεί μια μεταγραφή. Έπειτα για τους πράκτορες Υπάρχουν τα κριτήρια της FIFA που θέλουν να μειώνεται στο 3% η προμήθειά τους για τις μεταγραφές. Η προστασία των ανηλίκων. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε οι ανήλικοι και οι ανήλικες να προστατεύονται και στον αθλητισμό. δηλαδή ότι δεν θα χρησιμοποιούνται ανήλικα παιδιά σε αθλητικές δραστηριότητες και να προβλεφθεί μια κατώτατη ηλικία για τα πρωταθλήματα μεταξύ 16 και 18 ετών έτσι ώστε ένας αθλητικός σύλλογος που έχει αθλητικές δραστηριότητε στο εξωτερικό να πρέπει να μπορεί να αποδείξει ποια είναι η ηλικία των αθλητών του. Πρέπει επίσης να δούμε πώς αθλούνται οι ανήλικοι και οι ανήλικες. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες εξάσκηση επίσης των νεαρών αθλητριών. Το άρθρο 165 της Συνθήκης της Λισαβόνας λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει για να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές διαστάσεις του αθλητισμού. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ίσω πρέπει να προσθέσουμε ένα κεφάλαιο που θα είχε τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ταυτότητα του Αθλητισμού». Στόχο θα είχε να ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές αξίες και τα ιδεώδη μέσω του αθλητισμού. Θα ήθελα, παραδείγματι, να επικαλεστώ ένα ε, ιδιαίτερο άθλημα, μοναδικό, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται από μία, θα εκπροσωπείται από μία μόνο ομάδα και που θα ανακουγόταν και θα ακουγόταν ε, ο Ευρωπαϊκός ύμνος. Θα ήταν, αν θέλετε, το κορυφαίο ε, άθλημα. Κάθε Ευρωπαίος ε, πολίτης θα πρέπει να μπορεί να αποφελείται από τον αθλητισμό. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή μέρα του αθλητισμού. Θα ήταν η ευκαιρία για τη διοργάνωση συνεδρίων σχετικών και γεγονότων που συνδέουν τον αθλητισμό, για να μπορούν να μοιραστούν από κοινού το πάθος στον αθλητισμό. Θα μπορούσαμε σε συνέχεια βέβαια να οργανώσουμε και κάποιες ειδικέ εκδηλώσεις. Θα πρέπει στη συνέχεια να επιμείνουμε στη σημασία της ε, εξάπλωσης και της δημιουργίας ευρωπαϊκής πρωτεύουσα αθλητισμού. Θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα ευρωπαϊκό φεστιβάλ ε, αυτόχτονου αθλητισμού. Ε, επιμένω σε αυτό. Στα κράτη-μέλη και στις διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, ιδιαίτερα αθλήματα αποτελούν κομμάτι της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και αναγνωρίζονται και από την UNESCO. Θα πρέπει να εκπονήσουμε μια, ένα κατάλογο με όλα τα σχετικά αθλήματα και θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα ευρωπαϊκό σχετικό φεστιβάλ που θα ήταν αφιερωμένο στον τον αθλητισμό. Θα προτείνω επίσης τη δημιουργία ενός προγράμματος ευρωπαϊκού προγράμματος Εράσμου στον αθλητισμό που θα ήταν αφοσιωμένο στους νεαρούς ε, αθλητές και προπονητές θέτοντας κάποιους συγκεκριμένους στόχους που θα επέτρεπε στους ε, αθλητές να, να προπονούνται με διάφορους αθλητικούς ομίλους και στο εξωτερικό, να διευκολύνονται οι ενταλλαγές αθλητών στα διάφορα σχόλια, σχολεία δίνοντας δυνατότητα να μάθουν και μια ξένη γλώσσα, να ανακαλύψουν ένα καινούργιο πολιτισμό και να μάθουν και μια καινούργια μέθοδο ε, προπόνησης. Θα επέτρεπε επίσης τη διευκόλυνση ανταλλαγών μεταξύ ε, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο διαφόρων αθλητών. Οι διάφορες επίσης ευρωπαϊκές ομάδες που συμμετέχουν σε διεθνή πρωταθλήματα θα έπρεπε να προσθέσουν πέραν των εθνικών του συμβόλων και το ευρωπαϊκό, κάποιο ευρωπαϊκό σύμβολο. Έτσι λοιπόν, συνενώνοντας τις ομάδες μας, μπορούμε να δώσουμε ένα νέο άλμα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Ευχαριστώ εκτενέστατη η παρουσίαση. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο εν μια αλλά στον αθλητισμό χρειάζονται πολλές προτάσεις και πρωτοβουλίες και ο Σαντιάγκο τις είπε όλες. Ε, έχω κάποιους που έχουν δηλωθεί να μιλήσουν. Στη Γερμανία, σε ένα μεγάλο μόσφοντο κρατήδιο, γίνονται κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις και σκέφτηκα για τους ε, εκπαιδευτές ή τους προπονητές. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών είναι σημαντικότερη από ποτέ σήμερα. Έχουν μια τρομερή ευθύνη για τους νέους ανθρώπους και πολλά μπορούν να κάνουν για τη διπλή σταδιοδρομία, αθλητική και τη δεύτερη εάν έχουν το σχετικό προσανατολισμό και ετοιμασία. Και κάποιος μου είπε από την Ακαδημία, γιατί έχουμε μια μεγάλη Ακαδημία Αθλητισμού στην περιφέρειά μου, ότι δεν υπάρχει πτυχίο bachelor που να συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Στην Πολόνια υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το δίπλωμα bachelor ε, πρέπει να κάνουμε και το μάστερ, αλλιώ δεν γίνεται. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα μπορούσαμε στην ε, Ακαδημία να μπορεί να ολοκληρώνονται οι σπουδέ με το bachelor, δίνοντας έμφαση και στην αναγνώριση της εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι κάτι τέτοιο δυνατόν, γιατί όλο και περισσότερο νομίζω ότι θα είναι δυνατόν οι εκπαιδευτές που έρχονται σε επαφή με τους νέους να έχουν πιο καλά, ε, πιο στέρεες γνώσεις και αργότερα όταν δεν θα είναι πια εκπαιδευτές θα μπορούσαν ίσως με το πτυχίο αυτό να ασχοληθούν σε κάτι άλλο. Αυτά ήθελα να πω έχοντας ακούσει τις πολλές προτάσεις σου. Να προσθέσω δηλαδή και αυτή. Και τώρα ο κύριος Μπάλετερ που ξέρει το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, μιλώντας τα Ολλανδικά. Ε, θα, μιλήσω, είμαι σύντομος γιατί ο Σαντιάγκο είπε όλα τα βασικά σημεία. ο εισηγητή έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, Επομένω δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε όλε αυτέ τι φιλοδοξίε του. Υπάρχουν τεράστιε προσδοκίε οι οποίες ε, βασίζονται στην έκθεση αυτή. Έχουμε βέβαια κάπως περιορισμένες ε, δυνατότητες παρά τη συνθήκη Λισαβόνας, αλλά πρέπει να υποστηρίξουμε τις φιλοδογίες ε, και τη φιλόδοξη προσέγγιση του εισηγητή. Περιορίζουμε σε δύο σημεία, αφενός το θέμα αλληλεγγύης και αφετέρου κάποιες ε, απειλές που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός, για τις οποίες ανέφερε ο Σαντιάγκο. Το θέμα της αλληλεγγύης δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν μπορούμε παρά να επιμείνουμε πάντα πάνω στο θέμα αυτό στις διάφορες υπεύθυνε ε, ομοσπονδίες και οργανώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη. Ο Σαντιάγκο μιλήσατε για την συλλογικότητα σε ό,τι αφορά την αναμετάδοση, την πώληση των δικαιωμάτων αναμετάδοση αγώνων. Είναι σημαντικό αυτό για την UEFA και για τι Εθνικέ Ομοσπονδίε, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά και για άλλα αθλήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πολύ πιο αλληλέγγυη κατανομή των δικαιωμάτων αναμετάδοσης. Πρέπει να επιμείνουμε ώστε οι αθλητικοί όμιλοι να επενδύουν περισσότερο στους νέους. Έχουν γίνει σχετικά διαβήματα, Πιστεύω όμως ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις στις διευθύνουσε διευθύνουσες αρχές των διαφόρων ομίλων και ομοσπονδιών για να επενδύουν περισσότερο στους νέους. Και από αυτού του πεδίου συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει μια... Μηδενική... Πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την, ε, ε, το εμπόριο ανήλικων παικτών. Είναι παράδεκτο. Πρόσφατα λάβαμε κάποιες προφορίες σε ό,τι αφορά τις, ε, ε, τις ε, βαλτικές χώρες όπου μεταφέρονται νεαροί ποδοσφαιριστές 14-15 ετών οι οποίοι μεταφέρθηκαν που ήταν στις κάτω χώρες και που θέλουν τώρα να τους μεταφέρουν στην ε, πρώτη κατηγορία Εθνική Ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας. Υπάρχουν προπονητές, managers, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα της FIFA ε, μεταφοράς αγοραπολισίας πολιτών, εξε, ε, παικτών, συγγνώμη, καινούριο σύστημα και που συνδέεται με το σύστημα θέλω, των σχετικών managers των παικτών. Η FIFA έκανε μια νέα πρόταση για το καθεστώ αυτό, να μην εργάζονται μόνο με αυτούς που έχουν τη σχετική άδεια, αλλά με οποιονδήποτε θέλει να είναι διαμεσολαβητής, να έχει την αξιοδότηση να το πράξει, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, όπως είπε ο Σαντιάγκο προηγουμένω σε ό,τι αφορά τα ποσά τα οποία διακυβεύονται και τα οποία μεταφέρονται από τον έναν διάμεσο στον άλλον ή από μία αθλητική ομάδα στην άλλη. Επίσης, τίθεται κάποιος, κάποια αροφή για τους μισθούς, ε, για τις αμοιβές αυτών των ε, διαμεσολαβητών. Θα χρειαστεί βέβαια κάποιος χρόνος μέχρι το 2012 και το δεύτερο, και ολοκληρώνω με αυτό, είναι οι απειλέ οι οποίε βαρύνουν στον αθλητισμό. Μιλήσαμε για εδώ το πάρισμα, δεν θέλω να επανέλθω από αυτού οι διαδικασίες ε, κυρώσεων. Πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχει κάποια οργάνωση σχετική. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή θα πρέπει να γίνει μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Και τέλος, πριν από δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της επανεκλογής του, ο πρόεδρος Πλατινή έκανε ευρωπαϊκή έκκληση, ζητώντας από τα κράτη-μέλη και από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης να ορίσουν κάποιον ε, αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνο για την ε, δίωξη φαινομένων διαφθοράς ε, και στημένων αγώνων. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα αναφέρουμε στην έκθεση του κυρίου Φίσα. Ευχαριστώ. Κατ' εξαίρεση δίνω το λόγο στον κύριο Μπόρις ε, γιατί μετά πρέπει να πάει σε σημαντική ψηφοφορία σε άλλη επιτροπή και προηγείται λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, έχω ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Θα ήθελα λοιπόν καταχάσει να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή γιατί βλέπουμε εδώ όλες τις προκλήσεις ε, οι οποίες ε, αντιμετωπίζει ο αθλητισμός. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλοι οι αθλητικά γεγονότα που είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα πρέπει να έχουν πολύ πιο προωθημένα ευρωπαϊκά σύμβολα. Δεν θυμάμαι τις ευκαιρίες, αν θέλετε, και διάφορους αγώνες ποδοσφαίρου ή χάντμπολ ή άλλων που να έχουν ευρωπαϊκά σύμβολα. Εν πάση περιπτώσει τα σύμβολα αυτά δεν είναι ορατά. Αυτή η διάσταση είναι απόλυτα απούσα. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα αυτή, γιατί έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία μέσω των συνθήκων να το επιτύχουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των ε, νεαρών ε, αθλητών, οι, επαγγελματικές, οι επαγγελματικοί αθλητικοί όμιλοι, οι επαγγελματικές ομάδες θα πρέπει να υποστηρίξουν ακόμα περισσότερο και να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν τους αθλητές αυτούς. Όπως ξέρουμε, σε ό,τι αφορά πάρα πολυάριθμους τομείς, δεν έχουμε εντό εισαγωγικών πάρα πολλούς αθλητές εκτός Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε την ε, πληροφόρηση που θα επιτρέψει να βρεθούν, να βρίσκονται οι ταλαντούχοι αθλητές και να εντάσσονται σε επαγγελματικές ομάδες. Ορισμένες φορές σε κάποιες ομάδες το 90% των μελών μιας ομάδας ε, ε, είναι εκτός συγκεκριμένη περιοχής ή και εκτός χώρας ή και ακόμα εκτός χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, η επαγγελματική εκπαίδευση των αθλητών, που, αυτών που προσεγγίζουν, η επαγγελματική κατάρτιση των αθλητών που φτάνουν στο τέλος της διαδρομίας τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τα ευρωπαϊκά τα Ευρωπαϊκά Φόρουμ και τις Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς. Γιατί οι αθλητές που χαίρουν μεγάλους κύρους στη χώρα τους θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία κατάρτιση. Ορισμένες φορές δεν έχουν κατάρτιση για να γίνουν προπονητές, για παράδειγμα, ή καθηγητές φυσικής αγωγής. Ε, ή κάποιο συγκεκριμένο αθλήματο. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε τη δυνατότητα εκπαίδευση μεγάλου αριθμού επαγγελματιών αθλητών, ώστε στη συνέχεια να μπορούν να γίνουν με τη σειρά του καλοί προπονητέ, καλοί καθοδηγητέ τη νεολαία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά άτομα στο τέλο τη αεδρομία του χάνονται και είναι τελείω απελπισμένα. Ενώ αντίθετα θα μπορούσαν να είναι μεγάλο όφελο για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Η κυρία Κάμαρτ Εύερτ. Ευχαριστώ. Καταρχήν ένα θερμό ευχαριστώ στον εισηγητή που μας έδειξε άλλη μια φορά πόσο πολύπλευρο, πολυεπίπεδο είναι το θέμα αυτό. Για να έχουμε μια καλή έκθεση μετά την πρόταση της Προέδρου μας για την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Είναι σημαντικό το πρόβλημα και δεν πρέπει να περιορίζεται βέβαια στους εκπαιδευτές που θα εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες μόνο, γιατί ιδιαίτερα στους νέους έχουμε πολλούς που είναι ε, επίτιμοι ή μη επαγγελματίες και θα πρέπει να βρίσκουμε κάποιον που να γνωρίζει μεν πώς θα μάθει μπάσκετ ή βόλη στα παιδιά, αλλά κάποιον που να έχει και παιδαγωγικές ικανότητες, δεξιότητες, που πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει όταν ε, έρχονται σε επαφή με παιδιά σε ευαίσθητη ηλικία. Πρέπει λοιπόν να δούμε και το θέμα των μη επαγγελματιών εκπαιδευτών για τους νέους. Επίση, κάτι άλλο. Σε ένα σημείο η ανακοίνωση της Κομισιόν με απογοήτευσε λίγο, γιατί ήλπιζα ότι η ανακοίνωση αυτή θα διευκρίνιζε και κάποια νομικά ζητήματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό να τονίσουμε ότι η Κομισιόν αναδεικνύει τον ιδιαίτερο ρόλο του αθλητισμού, που λέει δηλαδή ότι δεν έχει, μόνο, έχει και οικονομική διάσταση, αλλά έχει και πολιτιστική διάσταση, διάσταση ολοκλήρωσης ο αθλητισμός. Αυτή η ιδιαίτερη θέση του αθλητισμού παρουσιάζεται μεν ως ορισμός μέσα στο κείμενο της Κομισιόν όταν μιλάμε για το δίκαιο του ανταγωνισμού, όταν μιλάμε για τις ρυθμίσεις και τις οδηγίες ε, για τις επιδοτήσεις. Λείπουν όμως κάποιες διευκρινήσεις ε, ή τονίζεται, τονίζονται ότι θα μπορεί να υπάρχει κάποια ε, εξαίρεση σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, αλλά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει επιτούτης να ε, ελέγχεται εάν χρειάζεται, αν θα πρέπει να γίνει η επιδότηση και αν είναι ε, επαγγελματική ή ε, επαγγελματικός ο σύλλογος ή όχι. θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά να ελέγχεται εάν υπάρχει σύγκρουση με το δίκαιο ανταγωνισμού. Είναι ασαφές το κείμενο. Θα πρέπει η Κομισιόν να προβεί στις απαραίτητες διευκρινήσεις, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα για τους αθλητικούς συλλόγους στην Ευρώπη και να μην φοβόμαστε κάθε φορά ότι θα υπάρξει παραβίαση της συνθήκης ενδεχομένως ε, λόγω της ε, παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού. Επίσης η Κομισιόν λέει ότι η κεντρική εμπορία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δεν θεωρείται να, ότι αφορά τον ανταγωνισμό όταν τα κονδύλια κατανέμονται με αλληλεγγύη και όχι μόνο μεταξύ των επαγγελματιών. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού και επιδοτήσεων, χρειάζεται πάντως σαφέστερη γλώσσα από την Κομισιόν και θα ήθελα να φροντίσει για μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τους αθλητικούς συλλόγους η Κομισιόν. Και επίσης κάτι άλλο που με απογοήτευσε λίγο είναι ότι εδώ με μεγάλη ομοφωνία στο Κοινοβούλιο ψηφίσαμε υπέρ ενό ενιαίου συστήματος μιας διαδικασίας για την χορήγηση της άδεια. Εδώ η Κομισιόν κάνει ένα βήμα πίσω. Θα πρέπει να ελεγχθεί αν λέει αν ε, χρειάζεται αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μήπως θα, μπορούσαν να συντονίσουν το θέμα μεταξύ τους οι αθλητικοί σύλλογοι. Αλλά στην UEFA που είναι μεγάλη αθλητική σύλλογη δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και μικροί σύλλογοι που δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό για να παρακολουθήσουν και να φτιάξουν τέτοια συστήματα διοδότησης τα οποία θα είναι και νομότυπα για να μην φοβούνται ότι ενδεχομένως θα υπάρξει κάποια σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη τόλμη από την, από, από την πλευρά της Κομισιόν και να δούμε και εμείς την έκθεση τι μπορούμε να προσθέσουμε εκτός από αυτά που είπε η Κομισιόν και τι δικαιούμεθα και τι είναι θεμητό να αναμένουμε από την Κομισιόν όταν πρόκειται για νομοθετική διαδικασία και μεγαλύτερη ασφάλεια νομική βεβαιότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά πρέπει να κοιτάω λίγο και το ρολόι, γιατί σύντομα θα έχουμε ψηφοφορίε στην Επιτροπή. Άρα ενδεχομένω θα χάσουμε την επόμενη σύγχυση που είμαι σκιώδη θα Το... Η Μέρι Μπόλη θα μπορούσε να το χειριστεί. Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, λοιπόν. Καταρχά να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Σαντιάγκο. Καταρχά, συγγνώμη, να τον συγχαρώ για την ε, πολύ καλή διοργάνωση μιας πολύ οικοδομητικής ακρόασης με πάρα πολλά μέλη τα οποία έχουν συνεισφέρει. Οι κύριες πτυχές εδώ είναι καταρχάς ότι σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνδίκης Λισαβόνας μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αθλητισμού και θα πρέπει να αξιολογήσουμε το τι συμβαίνει. Συμφωνώ με τον Σαντιάγκο ότι θα πρέπει να δούμε ότι θα υπάρχει προστιθέμενη αξία αντί απλώς ε, να επιχαίρουμε ότι συμβαίνει σε ατομικό ή σε εθνικό επίπεδο. Είναι πραγματική ευκαιρία να δημιουργηθεί μια πραγματική αίσθηση ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα στο αθλητισμό, αντί να έχουμε απλώς τις ε, εθνικιστικές, ε, εθνιστικές παραδόσεις που όπως πολύ συχνά έχετε ήδη επισημάνει. Αυτή είναι μια διάσταση, διάσταση που ανέφερε ο Σαντιάγκο, να οργανωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, η επιδίωξη διαφόρων επιτευγμάτων, αθλητικών επιτευγμάτων. Δεύτερον, ανεξαρτήτως χρηματοδότης που έχουμε στην Επιτροπή, θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση αντί να εμπλεκόμεθα σε ανταγωνισμούς που έχουν, που έχουν εμπλακεί διάφοροι αθλητικοί οργανισμοί. Θα πρέπει να το αποφύγουμε. Το όλο ζήτημα και έχει τονιστεί και στην ακρόαση σήμερα. Είναι οι δύο πτυχές στο θέμα. Είναι ο επαγγελματίας αθλητή και η σταδιοδρομία την οποία ακολουθεί συνέχεια, το της αθλητική σταδιοδρομία, αλλά υπάρχει και ο ρασιτέχνη αθλητή, του οποίου η σταδιοδρομία λειτουργεί εν παραλίλω με την αθλητική του ζωή. Πολλά λοιπόν έχουμε να προσθέσουμε στο τι συμβαίνει ήδη και ιδιαίτερα στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών, ώστε και οι μεν και οι δε να μπορούν να έχουν ε, επικερδί αν θέλετε, στα υδρομεία και να μπορούν να παρθούν στον περισσότερο. Ενώ στο ταυτόχρονα δεν θα, δεν θα παρεμποδίρονται στα διαδρομία του επαγγελματική που συχνά συμβαίνει. Είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο να δουλέψουμε. Κάτι άλλο που ανέφερε στην άφηση εδώ και πολύ σημαντικό είναι οι διάφοροι φορείς για την καταπολέμηση του ντόπινγκ. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά για να υπάρξει κάποια διαφάνεια και κάποια συνέπεια και συνοχή στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Συνολικά όμως νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει σωστά. Έχουμε αναγνωρίσει τα παιδεία στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε και να προσφέρουμε προς τη αξία. Και τέλος, ένα μέρος των βασικών ε, στόχων για το 2020 είναι να ενισχύσουμε και πάλι τη διαβίου μάθηση και εν παραλίλω μαζί με τη γραπτή διακήρυξη η οποία, την οποία έχουν υπερψηφίσει οι βουλευτές είναι και διαβίου φυσική δραστηριότητα. Διαβίου αθλητισμό και την ακρίβεια διαβίου φυσική δραστηριότητα, το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζουν περισσότερο, υγιέστεροι και ταυτόχρονα να μαθαίνουν ε, αν θέλετε, και διδακτικά, αλλά και στο τεφάλι φυσική δραστηριότητα. Πρέπει να λοιπόν την έννοια αυτή. Ευχαριστώ. Κυρία Νεύλα, Λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς και πρωτίστως. Νομίζω ότι επιτέλους αρχίζουμε να μιλάμε για τον αθλητισμό και σε αυτή την επιτροπή μπορούμε να προσεγγίσουμε το θέμα επαγγελματικά και όχι μόνο με γενικά συνέδρια, αλλά και κάνοντας κάτι συγκεκριμένο. Ο Σαντιάκο ήταν πραγματικά ενθουσιώδης για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Πολλά έχουν λεχθεί εδώ και αυτά που μας είπε η Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά. Η καταπολέμηση του ντόπινγκ είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ε, ταυτίζομαι με πάρα πολλές προτάσεις ε, που παρουσιάστηκαν εδώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάρει σαφή θέση σε πολλούς ε, οργανισμούς αθλητικούς και να καταπολεμήσει τον ντόπινγκ. Αυτό που δεν αναφέρθηκε εδώ είναι η συνεργασία των διαφόρων μειονοτικών ομάδων στις αθλητικές δραστηριότητε, γιατί η κοινωνική πτυχή του αθλητισμού και η συμπερίληψη στην κοινωνία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να τονιστεί αυτό. Πρέπει να υποστηρίξουμε πάρα πολλές ε, ε ομάδες που σε πολλές περιπτώσεις εξαιρούνται από πολλές δραστηριότητε. Είναι εξίσου σημαντικό να τονιστεί το θέμα και η πτυχή της ισότητας των φίλων, ενισχύοντας τη θέση των γυναικών σε αθλητικούς οργανισμούς θα ήθελα να δω περισσότερες ε, γυναίκες ε, διαιτητές, ε, ε, θεματοφύλακες και ορισμένε φορές εκεί που υπάρχουν άνδρες ε, διαιτητές δεν βλέπουμε να ιδιαίτερα για την ένταξη γυναικών γιατί πιστεύουν ότι οι γυναίκες μπορούν να έχουν προκατάληψη σχετικά. Είναι σημαντικό επίσης να καταπολεμηθεί και να, και να αποφεύγονται οι βίες σκηνές καταπολέμηση του χουλιγανισμού δηλαδή. Είπα κάτι αστείο. Κάποιες ομάδες ε, αναγκάστηκαν να καταβάλουν ε, πρόστιμα διότι οι οπαδοί τους έχουν προκαλέσει μεγάλες οικονομικές ζημιές σε γήπεδα. Είναι σημαντικό να καταπολεμηθεί η βία στους αθλητικούς χώρους. Τώρα, η κίνηση και η ανταλλαγή φοιτητών αθλητικών ακαδημιών. Πολύ σημαντικό να επεκταθεί το σχετικό πρόγραμμα έρεσμου ή ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Αν κάποιο έρχεται από, από, μια χώρα, ταξιδεύει σε μια άλλη, για εκπαιδευτικούς λόγους και θα θέλει ταυτόχρονα και να αθληθεί, θα πρέπει όντως να μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να ασκήσουμε περισσότερο αυτή την κινητικότητα και στους ε, αθλητές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, μόνο πολύ μεγάλοι ε, αθλητικοί όμιλοι, κατά κύριο λόγο ποδοσφαιρικές ομάδε χρηματοδοτώνται, ε, η FIFA έχει του πόρου. Υπάρχουν όμω και άλλα αθλήματα που σου δεν είναι τόσο δημοφιλή, αλλά χρειάζονται ε, οικονομική υποστήριξη. Είναι σημαντικό λοιπόν σαφέστα να διαθέσουμε κονδύλια για να υποστηρίξουμε και αθλητικού ομίλου, αθλητικέ ομάδε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ταιριάζει πολύ καλά με το, αυτό που έχουμε φέτος το Ευρωπαϊκό Έτος ε, Εθελοντισμού. Πολλοί εθελοντές προσφέρουν πάρα πολλά χωρίς καμία οικονομική αποζημίωση. Θα ήταν λοιπόν πολύ καλή ιδέα να τους δώσουμε κάποια κίνητρα, άλλου είδους κίνητρα. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες, ευρωπαϊκή ομάδα δεν υπάρχει. Μπορείτε να σκεφτείτε μια ενιαία ε, μία και μόνη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομάδα. Θα ήταν ενδιαφέρουσα ιδέα και ευχαριστώ να την υποστήριζα, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα επιλεγούν οι παίκτες σε μια τέτοια ομάδα. Και τέλος, αλλά εξίσου μεγάλη σημασία, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, ε την πρόθεση και την εγκατάσταση των αθλητών. Αθλητών. Έχω πολλούς φίλους, για παράδειγμα, παίκτες χόκεϊ, που μου λένε είμαι αθλητής, δεν χρειάζεται να πάω σε σχολή. Χρειαζόμαστε και να τονίσουμε περισσότερη επιπρόσθετη εκπαίδευση για αυτούς. Κάποια μέρα θα τελειώσει η επαγγελματική του διαδρομή η αθλητική και θα πρέπει να βρουν κάποια άλλη θέση στην κοινωνία. Δεν είναι κάθε αθλητής. Ε, Μπέκαμ για να βρει διέξοδο. Πρέπει να δοθούν λοιπόν κάποια εργασιακά ε, κίνητρα και να έχουν δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και μια φεμινίστρια ανάμεσά μας. Ένα μεγάλο θέμα που βάζεται πάντα είναι το θέμα των γυναικών πέρα από την ισότητα των φύλων, έτσι δυναμικά. Η κυρία Μποσκότ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών θα ήθελα να δηλώσω, να σχολιάσω την έκθεση αυτή γιατί θα ήθελα να συνεργαστούμε Ήδη υπάρχει μια ευρεία συνένεση ως προς την εισαγωγή της και την τύχη που θέλουμε να τις επιφυλάξουμε. Είναι σημαντικό να εγκριθεί, θα γίνει τελικά πολύ καλή έκθεση. Ιδιαίτερα από την άποψη που μας ενδιαφέρει εμάς, τις δημόσιες ελευθερίες δηλαδή. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα του ρατσισμού στον αθλητισμό που φυσικά θέλουμε να το καταπολεμήσουμε καθώς και τα ειστημένοι αγώνες και θέλουμε γενικά να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά όσο για το ντοπάρισμα. Εδώ πρόκειται για θέμα παραβίασης του ιδιωτικού χαρακτήρα Υπάρχει και το θέμα της συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων ως προς διαμεθοριακά εγκλήματα, αλλά επίσης, επίσης λέγω, το θέμα των διεθνών αθλητικών γεγονότων όπου πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων για να καταπολεμηθεί ο χουλιγκανισμός και ο τεντιμποϊσμός. Πρέπει να τονιστούν όλα αυτά πολύ περισσότερο. Αναμένω λοιπόν μεγαλύτερη συνεργασία με τον εισηγητή γιατί έχει περισσότερη εμπειρία από μένα. Σε όλα μέσα είναι η Λίμπε και στον αθλητισμό. Ε, ε δεν ξέρω, δεν πιστεύω να θέλουν να ζητήσουν να προσθεθεί κάτι και στο χάρτη θεμελιδών δικαιωμάτων γι' αυτό, αλλά πάντως καλό είναι να ασχολούνται πολύ. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε εισηγητή που δείχνει τέτοιο ενθουσιασμό για τον αθλητισμό. Σαντιάγκο, χαιρετίζω αυτό που είπες για την επικουρικότητα. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να σεβαστούμε την αυτονομία των αθλητικών ε, συλλόγων κλπ. Δεν είναι θέμα τι μπορεί να κάνει ο αθλητισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αντίστροφα. Και πρέπει να επικεντρωθούμε πού μπορεί η Ευρώπη να προσθέσει αξία και πού θα καταδειχθεί αυτό. Χαιρετίζω, Σαντιάγκο, τι ιδέε σου για τη συλλογή δεδομένων επίσης για όλα τα αθλήματα και καλό είναι να ενθαρρύνουμε τον αθλητισμό που προάγει την υγεία, καταργεί τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τώρα για τη χρηματοδότηση του αθλητισμού πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην παρέμβουμε υπερβολικά και να μειώσουμε τη χρηματοδότηση των αθλητικών συλλόγων που πουλώντας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να εξασφαλίσουν ε, κάποιους τοπικούς συλλόγους, να μην βλάψουμε δηλαδή τη χρηματοδοτική δομή που λειτουργεί ήδη. Πρέπει επίσης να δούμε καθαρά προσεκτικά τα ζητήματα των στοιχημάτων και να δούμε και το ζήτημα της ακαιρεότητας. Μην επικεντρωθούμε μόνο στον υψηλών επιδόσεων αθλητισμό, να δούμε και σε τοπικό επίπεδο τι μπορεί να γίνει. Εκεί ελπίζομαι να ε, καταφέρουμε πολλά αποκτώντας ε, μια αρμοδιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό. Από το στόμα σας εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα λόγια. Η κυρία Κώστα. Θεωρώ ότι η έκθεση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ευρύτατη και με πάθος που διέπει γενικά το διάγκο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και για το σύγχρονο μια άλλη πρωτοβουλία που μπορεί να παρουσιαστεί. Θα ήθελα να διαβάσω το τι έχει προκύψει. Ήθελα να πω κάποια πράγματα. Πρώτον, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά τον αθλητικό κόσμο θεωρήθηκε πέρα από τις ε, προβληματικές της ε, Λευκής Βίβλου που θα ανοίξει ευρύτερα το θέμα. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή θέλει μάλλον να επαναπροωθήσει πολύ πιο έντονα κάποια σημεία που η ανακοίνωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ πιο απαλή και ίσονος σημασίας. Κάτι το οποίο σημειώσαμε ήταν ότι η ανακοίνωση ε, συντάχθηκε ακούγοντας σχεδόν κατά αποκλειστικότητα τους σημαντικούς πρωταγωνιστές των επαγγελματικών ε, ε, οργανώσεων και του αθλητισμού αλλά ακούγοντας και λαμβάνοντας ελάχιστα υπόψη τις ε, τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη σύσταση των αθλητικών οργανώσεων. Υπάρχει δηλαδή, γι' αυτό και εκτιμώ ιδιαίτερα ότι Σαντιάκο ήθελε να τονίσει, αν θέλετε, μια προσέγγιση περισσότερο από τη βάση. Μια θεματική ενός, ε, αν θέλετε, δικαιώματος στην αθλητική δραστηριότητα που συμπληρώνει, αν θέλετε, και το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας γιατί είναι και θέμα κοινωνικής ένταξης, δημόσιας υγείας κλπ. Δεύτερον, νομίζω ότι χάνεται λίγο στην ανακοίνωση η αναγκαιότητα, η αναφορά, αν θέλετε, στην τοπική διάσταση. Δηλαδή, χρειάζεται και ένας ελάχιστος συντονισμός για να, που θα εγγυάται ότι όλοι οι πολίτες, ακόμα και στις τοπικές κοινότητες και όλες οι σχολικές μορφές θα έχουν και θα αναπτύσσουν κάθε αθλητισμό που συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Και μια έντονη ένταξη των ε, ε, εδαφικών και εθνικών πολιτικών έχει να κάνει το όχι μόνο αθλητισμό, αλλά και με τους σχολικούς θεσμούς, ε, με τους ε, πολυδομικούς οργανώσεις κλπ. Και στο θέμα των εγκαταστάσεων, ε, το θέμα της προσπέλασης εγκαταστάσεων αθλητικών που θα πρέπει να υπάρχουν παντού. Υπάρχουν τεράστιες ενσωροπίες στις χώρες μας και υπ' αυτή την έννοια πολλά πρέπει να γίνουν. Μια άλλη θεματική που θεωρώ είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί είναι τη δυνατότητα αθλητικής δραστηριότητα και την τρίτη, την τρίτη ηλικία. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Ένα δεύτερο ζήτημα για να συμπεριληφθούν και άλλα θέματα. Για τα υπόλοιπα ε, ε, συμφωνώ με αυτά σε ό,τι έλεξαν για τα δικαιώματα στον αθλητισμό. Το θέμα για τα διάφορα τίτλα, τίτλους, διπλώματα, πτυχία, αν θέλετε να πιο επαγγελματική χρειά του αθλητισμού. Αυτή η αναφορά που γίνεται και που τη συμμερίζομαι στο να γίνει καλύτερος ορισμός, ε, καλύτερος ορισμός ε, αντιστοιχίας σχετικών διπλωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μία από τις επιτυχίες που μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο και στα πλαίσια της Μπολών, ε, γιατί υπάρχουν διαφορετικά διπλώματα και το περιεχόμενο το εκπαιδευτικό είναι διαφορετικών επιπέδων και αναλαμβανωτικότητα και σε αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ένα άλλο σημείο, μένω λίγο αν θέλετε στην ουσία, γιατί η καταπολέμηση του ντόπινγκ δεν είναι μόνο ε, στα θέματα, αν θέλετε, του επαγγελματικού αθλητισμού, αλλά και στα γυμναστήρια. Υπάρχει τεράστιος κίνδυνος, αν θέλετε, και ιδιαίτερα στην υγεία των νεαρών παιδιών, των εφήβων, γιατί τα διάφορα αναβολικά, τα οποία είναι μορφή ντόπινγκ, διατίθενται σε καθημερινότητα, στην ε, στην καθημερινή ε, γυμναστική των παιδιών, σε οποιοδήποτε γυμναστήριο και με πυρολάξει του ελέγχου στα διάφορα ε, διατροφικά συμπληρώματα. Πρέπει λοιπόν να, να, το, να το προσέξουμε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα για τη δημιουργία, αν θέλετε, και την ε, ενίσχυση μια ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω του μέσω του αθλητισμού και μπορούμε να το δούμε και με τη θέση φυσικά του προγράμματο Εράσμου για τον αθλητισμό μια ευρωπαϊκή ομάδα, αν θέλετε, θα μπορούσε να ξεκινήσει ίσως, δεν ξέρω, ίσως με έναν αγώνα ποδοσφαιρικό μεταξύ Ευρωπαίων, ε, ε Ευρωπαίων ε, βουλευτών απέναντι, αν θέλετε, στους δημοσιογράφους. Το είδα κάτι παράδειγμα που να γίνεται στην Ιταλία, βέβαια, που υπήρχε, ήταν μάλλον ε, πολύ δύσκολη σχετική εμπειρία. Ή αντίστοιχα μπορεί να γίνει και με γυναική ομάδα είναι ένα αστείο αν θέλετε για να δείτε τι θα πούμε. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε κάποιο συμβολικό σημείο σε ό,τι αφορά και τις γυναίκες, αν θέλετε, την ευρωπαϊκή ταυτότητα του αθλητισμού. Είναι κάτι που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την πρωτοβουλία αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους υπάρχουν προβλήματα ίσως όχι στην υπερβολική προπόνηση των πολύ νέων σε ό,τι αφορά τις ε, αθλητικές δραστηριότητε, αλλά και τη δυνατότητά τους επιλογής ομάδας. Υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες σε διάφορες χώρες και χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία της ε, δυνατότητας και της ελευθερίας επιλογής ε, των ε, παιδιών και της οικογενειών τους απέναντι στις ομάδες και θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία συγκρίσιμα. Σε πάρα πολλές λίγες χώρες, στην Αγγλία ή αλλού, συλλέγονται στοιχεία σε ό,τι αφορά την αθλητική δραστηριότητα και την εξάπλωση των λεγόμενων, θέλετε, κινήσεων στα γυμναστήρια ή αλλού. Δηλαδή τα στοιχεία μόνο στα επίπεδα επαγγελματικών ομάδων. Πρέπει να γίνει λοιπόν πολύ πιο μεγάλη παρακολούθηση σε ό,τι αφορά τι πρακτικέ, όχι μόνο σε επίπεδο ε, πρωτοαθλητισμού ή σε επαγγελματικέ ομάδε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάγκο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, τα τελευταία... Ε, παρακολούθησα ιδιαίτερα την τελευταία, όντως ο τελευταίος ε, δεν είναι και κάπως άχαρο γιατί σχεδόν τα πάντα έχουν ειδηλεχθεί. Πολλοί ανέφεραν ήδη ένα πρόγραμμα Εράσμους σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό και ήθελα να ζητήσω από τον φίλο και συνάδελφο Σαντιάγκο να το προσέξει ιδιαίτερα. Ακούσαμε τον καθηγητή Καλούτσι που, έκανε, που έδωσαν διαπρίσιο λόγο πραγματικά και έδωσε ιδέες πραγματικά που μου έμειναν χαραγμένες στη μνήμη. Ε, συμμερίσουμε κάποιες ε, ιδέες. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε την φοιτητική οργάνωση Εράσμους που είχε τη γενική της συνέλευση την περασμένη εβδομάδα και εκεί ήταν παρόν και ο κύριος Παλσμίτ, Σμιτ, παλιός και νυν πρόεδρος της ε, Ουγγρικής Δημοκρατίας και πάνω από 800 Ευρωπαίοι φοιτητέ συμμετέσχουν, γιατί όλοι είχαν επωφεληθεί από τα προγράμματα ανταλλαγή φοιτητών ε, Εράσμου. Και όλοι αυτοί έδιναν, έδωσαν μια ευρωπαϊκή διάσταση και στι ευρωπαϊκέ αθλητικές δραστηριότητε και στην όλη θεματική. Σε προσκαλώ λοιπόν, Σαντιάγκο, να δεις, ε, αν θέλετε, και να εξετάσεις όλα αυτά τα ζητήματα σε πάθη περίπτωση θα έχεις την υποστήριξη μας για την εργασία αυτή την οποία εκτελείς. Και σε συγχαίρω. Ευχαριστούμε. Σκριτλέσκα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι προφέρατε ωραία το δύσκολο επίθετό μου. Δεν θα επαναλάβω όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαντιάγκο για το σχέδιο της έκθεσης. Τον συγχαίρω. Είναι αυθεντία μεγάλη στον αθλητισμό. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο σύστημα κυρώσεων για να καταπολεμήσουμε τη διαφορά στον αθλητισμό και η ό,τι αφορά τους μάνατζερ των επαγγελματιών και όσων ε, είναι υπεύθυνοι για τα στοιχήματα. Ε, θα πρέπει να επιλέξουμε ένα καταξιωμένο σύστημα. Τώρα, για τις γυναίκες. Ζητώ την κατανόησή σας, γιατί είμαι και στην Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας δεν είμαι φεμινίστρια, αλλά ε, είναι καλό να υπάρχει ίση μεταχείριση των δύο φίλων. Είναι σημαντικό στην έκθεση αυτή να αναφερθούμε και στις αποζημιώσεις, απολαβές των επαγγελματιών ε, αθλητών, γιατί υπάρχει εδώ, υπάρχουν διακρίσεις, γιατί οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο. Και ένα καλό παράδειγμα είναι ο μαραθώνιος, γιατί τα πριν των ανδρών συχνά είναι πολύ ψηλότερα από εκείνα των γυναικών. Τρίτη παρατήρηση. Η ηθαγένεια πολλές φορές θέλουν να αλλάξουν η ηθαγένεια οι παίκτες, οι αθλητές για να καλύψουν καλύτερα τη σταδιοδρομία τους, να την προωθήσουν και συχνά αποκτούν καινούρια ηθαγένεια. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε αυτή την πορεία πολλές φορές τους ε, αθλητές, γιατί συχνά με πολύ συνοπτικές διαδικασίες ε, αποκτούν τη νέα τους ε, ηθαγένεια. Κάποιος που αρχίζει ε, από την Πολωνία μπορεί να συμμετέχει στην Ορβηγία σε πρωταθλήματα. Θα πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ε, ποιος αθλητής μπορεί να πάει σε ποια χώρα με ποια ηθαγένεια. Ευχαριστώ. Και ο Μάρκος Τουρία, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ομολογώ ότι η εισήγηση του συναδέλφου Σαντιάγκο πραγματικά με εξέπληξε, γιατί ήταν πραγματικά εντελεχέστατη. Ήταν μια πραγματικά έξοχη εισήγηση, γιατί έβαλε το εθελοντικό σημείο, στοιχεία κατά του ντόπινγκ, την ε, κοινωνικό ρόλο αθλητισμού για την τρίτη ηλικία, τον, σαν τρόπο ζωής, ε, στη δημόσια υγεία, τα θέματα των κονδυλίων και το οικονομικό ζήτημα, στο οποίο θα επανέλθουμε βέβαια θα έχουμε δεχτούμε την ε, Επίτροπο όταν μιλήσουμε και κάποιε πτυχέ για το πρόγραμμα Εράζου, τον αθλητισμό κλπ. Όπω είπαν ήδη και άλλοι συνάδελφοι, ο ρόλο μα είναι αυτός να καθορίσουμε μια προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι εθνικέ πολιτικέ αθλητισμού και τονίζω την ε, σημασία του να καταρτιστούν και να παγιωθούν κάποιοι κανόνες ε, συμπεριφοράς, το ρόλο της UEFA, της FIFA και τόσων άλλων. Η προσοχή μας λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στον βασικό αθλητισμό, αθλητισμό ε, αν θέλετε να δοθεί ε, δύναμη, όθηση και κίνητρα για να εξαπλωθεί ο αθλητισμός στους αθλητικές, σε επίπεδο ε, εθελοντισμού, σε επίπεδο βάσης, που θα πρέπει να είναι έντονο στην κοινωνία μα. Κοιτάζοντα ιδιαίτερα τον αθλητισμό στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, ω αφενό μεν ω ένα στοιχείο εκπαίδευση, αλλά και μια αθλητική δραστηριότητα, σκεφτείτε το πώ γίνεται στι ΗΠΑ, πόσα επενδύουν στον αθλητισμό, ακριβώ σε επίπεδο σχολείων, κολεγίων και πανεπιστημίων. Νομίζω είναι σημαντικό να πρηματοδοτήσουμε τον αθλητισμό σαν ένα στοιχείο συνοχή στι χώρε μα, στι 27 χώρε, και ω και ένα επίπεδο και ένα στοιχείο διασυνοριακού διαλόγου και ένα στοιχείο, όπως είπε προηγουμένως ε, συνάδελφος, ε, διαμόρφωσης, αν θέλετε, ευρωπαϊκής ταυτότητας. Να βοηθήσουμε επίσης τις χώρες μας να αναπτύξουν αθλητικές δομές γιατί εκεί που υπάρχουν καλύτερε αθλητικές εγκαταστήσει και υπάρχει τέτοια δομή και το περιβάλλον είναι καλύτερο, το δέχεται το περιβάλλον θετικά, αναπτύσσεται κανείς καλύτερα, υπάρχουν καλύτερες δομές. Βοηθά λοιπόν ο αθλητισμό τις ε, περιοχές μας να βελτιώσουν τι αθλητικές δραστηριότητε και αντίστοιχα αναπτύσσεται πολύ καλύτερη τοπική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε και την διαρθρωτική πολιτική και μήπως και αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Γιατί δεν έχουμε ατελείωτα κονδύλια στον προϋπολογισμό. Η Κομισιόν, ο κύριος Πέντρο Βελάσκεθ Φερνάντεθ, που είναι επικεφαλής ε, της Μονάδας για τον Αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Φίσα τον εισηγητή για την εξαιρετική παρουσίαση. Και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την έκθεση όπου αναφέρονται όλες οι βάσεις που χρησιμεύσαν για το έγγραφο της Κομισιόν. Ε, λάβαμε υπόψη τις ιδέες ε, που ανέφερε ο κύριος Φίσας ε, και που ε, σε μεγάλο βαθμό συμβιβάζονται με την πρωτοβουλία της Κομισιόν και αυτό το σημειώνουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στα νέα, στο νέο κεφάλαιο, για το νέο κεφάλαιο, την ευρωπαϊκή ταυτότητα στον αθλητισμό που ανέφερε ο κύριος ε, Φίσας. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα την παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα για τις ιδέες του κυρίου Φίσας, το σημαντικό, με τα σημαντικότερα συμφωνούμε για την, την επικουρικότητα, την αυτονομία που είναι απαραίτητα. Η Κομισιόν τα αναγνωρίζει αυτά στο εγγραφό της. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχουν λιγότερες χώρες στον κόσμο στις οποίες ε, υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία στον αθλητισμό από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει την ίδια αυτονομία επίσης όπως σε εθνικό επίπεδο ο αθλητισμό και πρέπει αυτό να μας κάνει περήφανου. Τώρα κάποια πιο επίκαιρα στοιχεία. Εδώ εκφράστηκε η θεμητή ανησυχία που την σημεριζόμεθα δηλαδή η προαγωγή της σωματικής υγείας μέσα από την εξάπλωση του αθλητισμού. Αυτό είναι θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ε, δουλεύουμε. Ε, σύντομα θα δημοσιευτούν και τα αποτελέσματα μιας μελέτης για τις ε, χρηματοδοτικές κινήσεις στον αθλητισμό για τον ευρύτερο πληθυσμό θα πάρουμε στοιχεία από τους 27 για τη χρηματοδότηση του μαζικού αθλητισμού, ε, ποια, ποιο είναι το ποσοστό των ιδιωτών. Νομίζω ότι και αυτό θα βοηθήσει στο έργο του Κοινοβουλίου. Ο επαγγελματικός αθλητισμός και εδώ εργαζόμεθα. Επίσης θα γίνει σύντομα μία μελέτη σε σχέση με τις ε, ε, αποσπάσεις ή μεταφορές ε, αθλητών. Επίσης θα γίνει μια διάσκεψη με μεγάλους συλλόγους ε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό θα γίνει τέλος του χρόνου, το Νοέμβρη συγκεκριμένα. Επίσης λαμβάνω υπόψη μου το γεγονός ότι υπάρχει πρόθεση στην έκθεση να αναφερθεί και μια έκκληση σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση των αθλητών ηλικίας 16 με 18 ετών. Ζητείται ο περιορισμός της ελευθερίας διακίνησής τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό που πρέπει να το μελετήσουμε σε βάθος, γιατί σε τελευταία ανάλυση ε, θα πρέπει να δούμε τι θα πούμε σε ένα νέο. Δεν μπορούμε να του πούμε ότι μπορεί να εργάζεται οπουδήποτε εκτός από τον αθλητισμό. Για να το κάνουμε αυτό χρειάζονται πολύ στέρεα επιχειρήματα για να προβούμε στις απαραίτητες ρυθμίσεις. Επίσης κάνουμε διάλογο με την UEFA και την FIFA, διότι μας προσήγγισαν για να συζητήσουμε το θέμα της ελεύθερης διακίνησης. Θέλουν να απαγορευτεί για αθλητές 16-18 ετών. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι τα κίνητρα αυτών των ετοιμάτων. Επίσης κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, σχετικά με τους ε, στημένους αγώνες. Θα κάνουμε μια μελέτη επίσης προς το τέλος του χρόνου για να δούμε πώς θα καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό. Εκεί θα γίνει ανάλυση για κάθε κράτος μέλος και θα γίνει και ένας απολογισμός. Ποια είναι η θέση του αθλητισμού, και ποια είναι η σχέση του με το ποινικό δίκαιο. Αν υπάρχει διαφθορά στον αθλητισμό, για παράδειγμα, προβλέπεται, είναι ποινικό αδίκημα, ε, γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη συμβαίνει αυτό, σε άλλα όχι. Οπότε πρέπει να έχουμε μια συνολικότερη εποπτεία της κατάστασης του 27. Για το ντόπινγκ συμφωνούμε με αυτά που είπατε και εργαζόμεθα πάνω σε αυτό το θέμα ούτως ώστε να προσχωρήσουμε ε, στην σύμβαση κατά του ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, ε, το ντόπινγκ στο μαζικό αθλητισμό είναι προτεραιότητα για μας και γι' αυτό σε μια ανακοίνωσή μας τονίζουμε ε, ότι είναι σημαντικό να καταπολεμήσουμε το εμπόριο με ουσίες ντόπινγκ. Αυτά. Ε, το μόνο που μένει είναι να επαναλάβω ξανά τις ευχαριστίες μου για το εξαιρετικό έργο του Κοινοβουλίου και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε και στο μέλλον μαζί σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βελάσκεφ Χερνάντετ και ο κύριος Φίσας που έχει τον τελευταίο λόγο. Σαντιάγκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ ευχαριστώντας τους πάντες, όλους τους συναδέλφους για τα πολύ ευγενικά λόγια που είχαν για την ε, έκθεση αυτή. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας. Ε, σημείωσα τις ε, διάφορες ε, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας που λίγος πολύ φαίνεται να γίνονται προς την ίδια κατεύθυνση που έχω θέσει. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο όρια. Η επικουρικότητα αφενός, πρέπει δηλαδή να αποδεχθούμε ότι οι αρμοδιότητες σε σχέση με τον αθλητισμό εξακολουθούν βέβαια να είναι το κρατών μελών και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, και σε περιφέρειες, όπως σημαίνει στην Ισπανία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, ίσως και σε άλλες χώρες. Και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο όριο, που είναι οι αθλητικές ομοσπονδίες. Αθλητικές ομοσπονδίες οι οποίες είναι ελεύθερες να οργανωθούν κατά το δοκούν και ούτε και αυτό δεν θα θέλαμε να το αλλάξουμε. Όμως βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Η επικουρικότητα λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση. Πρέπει να μελετήσουμε κάθε πιθανή εξαίρεση και να καθορίσουμε κατά πόσον ε, υπάρχει συμμόρφωση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιτρέψτε μου να αναφέρω κάποια σημεία. Οι Ντόρις και άλλοι ανέφθηκαν ε, στην κατάρτιση για τους ε, προπονητές. Ε, υπάρχουν διάφορες τύπου, διάφορο τύπου προπονητές, αν θέλετε. Υπάρχουν εθελοντές που επίσης πρέπει να καταρτιστούν. Γιατί αν δεν είναι εκπαιδευμένοι μπορούν να προκαλέσουν και κακούς αθλητές. Υπάρχουν προπονητές, ε, ε, εκπαιδευτές, αν θέλετε, γενική τη γενική τη αλλά υπάρχουν πιο συγκεκριμένα τεχνικοί του αθλητισμού προπονητές που μπορεί να έχουν κάποια προσόντα και κάποιο δίπλωμα από κάποιο αντίστοιχο κολέγιο της χώρας τους και υπάρχουν και άλλοι εκπαιδευτές εξειδικευμένοι προπονητές για κάθε άθλημα. Οπότε εκεί ενδεχομένως θα μπορούσε να αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, κάποιο δίπλωμα τα διάφορα προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχουν ε, για κάθε έθλημα, ώστε κάποιος ο οποίος έχει αν θέλετε κάποιο συγκεκριμένο προσόν, κάποιο δίπλωμα στη Γερμανία να γνωρίζεται αντίστοιχα συμπλήν ε, κάτι επιπρόσθετο σε άλλη χώρα. Συμφωνώ επίση ό,τι αφορά την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αναμετάδοση. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο αυτό που αφορά στην Ευρώπη γιατί κάποιοι ε, αθλητικοί όμιλοι ε, δεν έχουν το δικαίωμα και δεν μπορούν να διαθέσουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα να μετάδουν στον αγώνα τους όπως ε, επιθυμούν. Είναι μία από τις ιδιαιτερότητες οι οποίες, αν θέλετε, ίσως είναι λογικές και πρέπει να γίνουν αποδεκτές για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Αθλητικού Μήλου της Βαρκελόνης, για παράδειγμα, της Βαρσελώνα, αποδέχεται ότι πρέπει να υπάρχει κάποια συμβιβαστική συμφωνία επί του θέματος. Τώρα, η στρατολόγηση και η μεταφορά και το εμπόριο, αν θέλετε, οι μεταγραφές ανήλικων αθλητών. Προφανώς ε, το, 10, το όριο των 18 ε, ετών, αν θέλετε, εξασφαλίζει αυτό το θέμα. Αλλά οι Γάλλοι έχουν πολύ έντονη θέση. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνει αυτό που λέει η Γαλλία ή η FIFA, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ε, του θέματος και θα πρέπει να, σας, να γίνει σεβαστό. Η προστασία των ανηλίκων είναι θεμελιώδης σημασία για μένα. Μιλήσαμε περί γυμναστικής και δινεαρών γυμναστριών που πολύ συχνά εμποδίζονται στην ε, φυσική τους ανάπτυξη λόγω των πρακτικών που εφαρμόζονται στην ε, προπόνησή τους. Αυτό είναι παράδεκτο. Πρέπει να υπάρχει προστασία των λύκων στις μεταγραφές τους. Όλα αυτά είναι αλλοσυνδεόμενα ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την αρμόνιση των ε, πιθανών κυρώσεων, Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε εκτενώς. Νομίζω ότι το, το, το αθλητικό δικαστήριο στην Ελβετία θα πρέπει να έχει κάποιο ισοδύναμο στην Ευρώπη, όπως έχει η Αυστραλία ή η Γιατί ο ελβετικός, το ελβετικό δίκαιο είναι πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Ίσως εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή σημαία και τα ευρωπαϊκά σύμβολα σε αγώνες, συμφωνώ επίσης. Το, το τι συμβαίνει στους αθλητές στο πέρας στα διαδρομία τους είναι επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν το ανέφερα προηγουμένως, αλλά Σκέφτομαι το γιατί οι επαγγελματίες αθλητές δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση. Ίσως δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο μισθό με το πέρας της αθλητικής αεροδρομίας. Και συμφωνώ με την Doris για, την, για τους ε, ε, προπονητές όπως είπαμε. Τώρα κάτι που θέλω να πω σχετικά με το στοίχημα, ε, τα αθλητικά στοιχήματα. Υπάρχει κάποια σχετική πράσινη στην Παγνία για το θέμα του στοιχήματο, Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα των ε, αθλητικών οργανώσεων, οι ίδιοι οι, οι διοργανωτές να επιλέγουν το στοιχηματισμό, τον οργανισμό, αν θέλετε, στοιχηματισμό που είναι καλής πίστης. επί της ε, ουσίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι στο δυνατόν οι διάφορες ομοσπονδίες να επιδεικνύουν αλληλεγγύα, κάθε αλληλεγγύη, δηλαδή η κάθε ομοσπονδία να εντάσσεται σε ευρύτερη συνομοσπονδία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, γυναίκες αθλητρίες, δεν πρέπει να βάλουμε, μάλλον όχι αθλητρίες, αλλά σε διοικητικά ε, πόστα, σε ομοσπονδίες ε, δεν θα πρέπει να είναι ένα θέμα ποσοστώσεων, αλλά θα πρέπει να λειτουργούν με ισότιμους όρους όπως στους άντρες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει προώθηση και προαγωγή του αθλητισμού στις γυναίκες. Υπάρχει και το θέμα χρηματοδότησης των ε, διορθωτικών ταμείων. Ακούσαμε περί επικουρικότητας, ναι, αλλά δεν μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εκλειφθούμε ότι βοηθάμε με μονομένους ε, ομίλους ή ομοσπονδίες. Αυτό πρέπει να το κάνουν πόλεις, αν θέλετε, οι περιφέρειες. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε ευρύτερες κλίμακας ε, ε, προγράμματα, όπως ένα πρόγραμμα Εράσμους για τον αθλητισμό. Και σε ό,τι αφορά θέματα δομής. Γιατί ο πολιτισμός μπορεί να τύχει κοινοτική σωματοδότηση και όχι ο αθλητισμός. Πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριληφθεί και ο αθλητισμός και δύο σχολικός τεχνικός στα πεδία των διαρθρωτικών πολιτικών που εκπονεί και εφαρμόζει. Η κυρία Πόρκλουτ είπε κάτι περί ρατσισμού, ναι, η καταπολέμηση του ρατσισμού και ε, της ε, ομοφιλοφοβίας μέσω αθλητισμού και βέβαια είναι αναπαράδεκτες ε, οι θέσεις αυτές. Τώρα, τα στημένα παιχνίδια σημαντικό το θέμα. Αν αναγνωρίσουμε όμως αυτή την ελευθερία στους ε, οργανωτές διαφόρων αθλητικών ε, αγώνων Ίσως ε, σε αυτά τα πλαίσια μπορεί, εκεί, εκεί αν θέλετε βρίσκεται και το πρόβλημα. Τώρα, το ντόπινγκ είναι σαν τα ναρκωτικά. Πρέπει να το προσεγγίσουμε αντίστοιχα με το πώς αντιμετωπίζουμε το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Χρειάζεται διεθνή συνεργασία και πρέπει προφανώς να διώκονται οι θρέμποροι ουσιών ντόπινγκ. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Αισθανόμαι πολύ Ευρωπαίο σήμερα. Όντως πρέπει να υποστηρίξουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα Εράσμους. Και σας διαβεβαιώ, η επικουρικότητα κατ' εμέ είναι ζωτική σημασίας. Δεν είπα ότι πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκές ομάδες για διάφορα αθλήματα. Δεν σε αυτό καθόλου κάτι τέτοιο. Αλλά όλοι έχουν, ας πούμε, κάποιο περιβραχιόνιο με την σημαία της χώρας τους όταν ε, αγωνιζόμαστε σε εθνικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και μια μικρή ευρωπαϊκή σημαία, ευρωπαϊκό σύμβολο. Βέβαια, εξαρτάται από τις ομοσπονδίες εμφάσεις θέλουν να κάνουν, αλλά είναι μια δυνατότητα. Θα έπρεπε να πούμε ότι θέλουμε, και να το πούμε στην Επιτροπή, ότι θέλουμε να είναι η γνωμοδότησή μας συμπληρωματική στην ε, σχετική ανακοίνωση. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε. Πρέπει να εφαρμοστούν, αν θέλετε, οι αρχές ε, της χρηστής διακυβέρνησης και σε περιφερειακό επίπεδο. Ακούσαμε περί το παρίσματος. Κατά κλείδι γίνονται ιατρικές εξετάσεις και ιατρική έλεγχη στο επαγγελματικό επίπεδο αθλητισμού, όχι στο τοπικό αριστεχνικό επίπεδο. Και πρέπει να δούμε τι κανόνες ισχύουν και στο βασικό επίπεδο αθλητισμού. Δεν είναι δίκαιο για κάποιο όμιλο για κάποια αθλητική ομάδα η οποία έχει τύχει πολύ μεγάλη χρηματοδότηση ε, να χάνουν ένα ταλέντο το, στο οποίο έχουν επενδύσει λόγω μεταγραφή ή λόγω κάποιε απώλειε. Κάποιε συγκεκριμένε προδιαγραφέ πρέπει να τηρούνται. Ανέφερα, αναφέρθηκε το πρόγραμμα Εράσμου. Η Τζοάννα μίλησε για κυρώσει σε περίπτωση διαφθορά. Πρέπει να τηρουνται αναφερθηκε το κατά πόσον μπορούμε να επιτύχουμε σχετική συμφωνία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Οι γυναίκες αναφέρθηκε αυτό, συμμετοχή των γυναικών και στα διοικητικά πόστα, στον αθλητισμό, στι αθλητικές ομοσπονδίε. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό ξέρω από του οργανωτέ, από τους φορείς. Εάν θέλουν να πληρώνουν περισσότερο του ε, επίσης τους άντρε αθλητές, ε, στην ενισότητα δηλαδή ε, απολαβών αντρών και γυναικών αθλητών, δεν μπορούμε να του ξαναγκάσουμε να μην το κάνουν. Ορισμένες φορές πρέπει να σκεφτούμε ναι, ε, παραπάνω σε ό,τι αφορά τις ε, διεθνείς μεταγραφές αθλητών. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τον βασικό αθλητισμό, αθλητισμό στην βάση, αναφέρθηκε. Θέλω να πω στον Μάρκο ότι ο πανεπιστημιακός αθλητισμός είναι σημαντικός, όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στη ΣΥΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη. Ο, αθλητικό, ο εραστηνικός αθλητισμός ε, ανθεί σε πανε, πανεπιστημιακό επίπεδο στις ΗΠΑ, ενώ εδώ στην Ευρώπη ανθεί σε επίπεδο ομοσπονδιών. Υπάρχει λοιπόν ε, θεμελιώδης ε, δομική διαφορά. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Και εξακολουθώ έχω κι άλλο να πω, ε. Μακάρι να το χρόνο. Δεν είναι η τελευταία φορά που τα συζητάμε όλα αυτά. Έχεις χρόνο, γιατί τον ε, Ιούλιο θα φέρει το σχέδιο. Μέχρι τότε θα κάνεις πολλές διαβουλεύσεις με πολλούς και η ψηφοφορία θα γίνει αρχές Οκτωβρίου. Οπότε ας δώσουμε χρόνο για όλα αυτά. Μόνο μην μπερδεύεις το Εράσμους με το... Μην μπερδεύεις το Εράσμους. Κάθε ε, φοιτητής ε, ε, της Ακαδημίας του Αθλητισμού μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα Εράσμους. Εσείς και άλλοι θέλουν την ιδέα του Εράσμους να την διευρύνεις σε ένα άλλο επίπεδο για να μην νομίζει κανείς ότι δεν μπορεί κανείς να πάει όταν σπουδάζει σε μια ε, ε, Ακαδημία Φυσικής Αγωγής ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα Εράσμους αυτό θα ήταν η λάθος εντύπωση γιατί μπορεί Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Σαντιάγκο, καλή επιτυχία στη δουλειά σου και προχωρούμε τώρα ε, στο επόμενο. Η κυρία Χάνιουελ για την αντιμετώπιση της προώρης εγκατάλειψης του σχολείου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. Πρόσφατα είχα γράψει μια έκθεση για τα πρώτα χρόνια της παιδείας και είναι καλό να μπορεί κανείς να δει το πράγμα και από την άλλη άκρη. Η πρώην κατάληψη του σχολείου είναι από τι μεγαλύτερε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε στην παιδεία. Το 2009 πάνω από 6 εκατομμύρια νέων έφυγαν από τα σχολεία και την παιδεία χωρίς να έχουν φτάσει μέχρι το απολυτήριο και 17% δεν τελείωσαν ούτε το δημοτικό. Και σχεδόν το 50% όσων εγκατέλειψαν το σχολείο παρέμειναν άνεργοι οι χώρες μέλη είχαν δεχτεί να μειωθεί σε λιγότερο από 10% ο αριθμός όσων φεύγουν ε, πρώιμα από τα σχολεία μέχρι το 2010, αλλά μέχρι τώρα μόνο 7 χώρες μέλη έχουν πετύχει το στόχο αυτόν. Τον Ιούνιο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε εκφράσει τον στόχο αυτό και είπε ότι αυτό το 10% μέχρι το 2020 αυτή τη φορά θα ήταν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής του 2020. Συμφωνώ βεβαίω με τη στρατηγική αυτή, θα ήθελα και να ενδυναμωθεί με την έκθεσή μου. Γιατί είναι τόσο σημαντικός λοιπόν αυτός ο στόχος, εκτό από τα τρομερά στατιστικά στοιχεία που ανέφερα, πρέπει να γνωρίζουμε και σε τι οδηγεί η πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου. Απαγορεύει τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την μάθηση. Και γι' αυτό αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ανεργία και την ανέχεια. Είναι άμεση η σύνδεση μεταξύ πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου και ανεχίας και πτωχίας και ανεργίας. Η, τα μακροπρόθεσμα ωφέλη για την κοινωνία αφορούν φυσικά την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εργατικό δυναμικό. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει αν μεγάλοι αριθμοί νέων φεύγουν από τα σχολεία πριν να πάρουν τα πτυχία τους ή τα απολυτήριά τους. Επίσης υπάρχει και κάτι πιο προσωπικό. Τα αποτελέσματα της πρώτης εγκατάλειψης του σχολείου αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων. Αυξάνουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και επομένω μειώνονται οι ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά στην υπόλοιπη ζωή τους και άρα το πρόβλημα της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου είναι πρόβλημα που αφορά πολλές γενναίες, όχι μόνο μία. Ποιος είναι ο λόγος της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. Προφανώς υπάρχουν ατομικές, ατομικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα παιδείας οι μεγαλύτεροι αριθμοί των προώρος εγκαταλειψάντων είναι από φτωχέ οικογένειες. Ή είναι παιδιά με γονείς χαμηλής εκπαίδευσης από φτωχέ οικογένειες, επαναλαμβάνω, με, καμιά φορά με αναπηρίες πνευματικές ή σωματικές που χρειάζονται ειδικέ ε, εκπαιδευτικές ανάγκες και μετανάστες, άλλα μέλη μειονοτήτων. Η εκπαίδευση και η παιδεία σε ολόκληρη την Ευρώπη πολλές φορές δεν χορηγεί καμία δυνατότητα υποστήριξης των μαθητών μπροστά σε τέτοιες δυσκολίες. Είναι βέβαια δεν είναι εύκολο να οργανωθεί κάτι τέτοιο και η πρώην κατάληψη του σχολείου γίνεται και θέμα φίλων τελικά γιατί περισσότερα αγόρια φεύγουν από το σχολείο προώρα παρά κορίτσια. 60% των εγκαταλειπώντων είναι αγόρια. 80 μάλλον. Τώρα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόορη αυτή εγκατάλειψη. Η Κομισιόν έγραψε μία ανακοίνωση όπου εξετάζει τρεις παράγοντες που πρέπει νομίζω και εμείς να δεχτούμε ως Επιτροπή. Πρόληψη, παρέμβαση και αυτό που λένε αντιστάθμιση εκείνη που φαντάζομαι σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για όσους τις έχουν χάσει από το σχολείο. Η πρόληψη σημαίνει πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου γιατί αυτό συνδέεται άμεσα με γιατί υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ καλής ποιότητος ε, από την προσχολική ηλικία ήδη παιδείας με την συνέχιση των σπουδών μέχρι το απολυτήριο. Επίσης, πρέπει να υπάρχει συστηματική γλωσσική στήριξη για παιδιά μεταναστών, πράγμα το οποίο δεν γίνεται πάντα όπως θα έπρεπε, και η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και της πρόσβασης σε αυτήν είναι σημαντικός παράγοντας, ώστε οι μαθητές και φοιτητές να μπορούν πιο εύκολα, αν συναντήσουν δυσκολίες, να ακολουθήσουν επαγγελματική κατάρτιση. Η παρέμβαση τώρα. Υπάρχει θετική παρέμβαση που μπορεί να γίνει, όπως η αντιμετώπιση των δυσκολιών από μικρή, από νεανική ηλικία, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ιδιαίτερα συνεννόησης με τους γονείς, δικτύωση με επαγγελματίες εκτός σχολείου που έχουν πρόσβαση σε δίκτυα στήριξης, προσωπικά συστήματα στήριξης της μάθησης και καλύτερη σύνδαση των δυνάμεων της αγοράς στον καθορισμό της των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης των νέων έτσι ώστε όσοι έχουν τον πειρασμό να φύγουν από το σχολείο να μπορούν να έχουν μια εναλλακτική επαγγελματική κατάρτιση. Τώρα η αντιστάθμιση και η δεύτερη ευκαιρία θα έπρεπε να δώσει νέες ευκαιρίες σε εκπαίδευση για όσους έχουν φύγει από το σχολείο ήδη. Να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία ώστε αυτό συνδέεται με όλη την ιδέα της διαβίου μαθήσεως. Ότι δηλαδή αφού πάρει κανείς το απολυτήριό του δεν τελειώνει η απαραίτητος η εκπαίδευσή του. Σε ενωσιακό επίπεδο νομίζω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε τη σημασία που έχει μεγαλύτερη συνεργασία. Μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα για τη στήριξη των χωρών μελών ώστε να εφαρμόσουν αποτελεσματικά εθνικά προγράμματα κατά της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. για να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια ως υποδείγματα Υπάρχει η ανακοίνωση, η δήλωση που αφορά την ε, σχολική εκπαίδευση από την αρχή ήδη της και επομένως ο καλύτερος συντονισμός θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι θα βρεθούν τα καταλληλότερα μέτρα για να αντιμετωπιστεί από τα κράτη-μέλη το πρόβλημα μέσω της εγκαθίδρυσης μηχανισμών που να εγγυώνται λίγο πολύ ότι δεν θα συμβαίνει τέτοια εγκατάλειψη πρόωρα του σχολείου και από τους εκπαιδευόμενους και από τους εκπαιδευτάς και εκπαιδευτρίας. Επίσης, πρέπει να επικεντρωθούμε στους ίδιους τους μαθητές και φοιτητές η πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου είναι πολύπλοκο φαινόμενο και πρέπει να δούμε καταρχάς ποιο είναι το κύριο συμφέρον του ατόμου και του ανθρώπου και του προσώπου. Πρέπει να εξετάσουμε πρώτα τα άτομα ή πρόσωπα για να Είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να μειωθεί ο αριθμός των ε, προώρως εγκαταλειπώντων τα σχολεία ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος του 10% μέχρι το 2020. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη συζήτηση και παρακολούθησε την έκθεση για την προώρη εγκατάλειψη σχολείου. Είναι πολύ δυσεπίλητο και δύσκολο θέμα και είναι σημαντικό να κάνουμε το δυνατόν για να μειώσουμε το φαινόμενο αυτό. Θέλω λίγο εξορροπώντας το θέμα αυτό να πω ότι δεν είναι πάντα κακό το ότι πολλοί φεύγουν γνωρίσω από το σχολείο. Πολλοί θέλουν να φύγουν για να μπουν σε επαγγελματική κατάρτιση ή γιατί έχουν κάποιες ε, ε, χειρονακτικές δεξιότητες που μπορούν να τις αναπτύξουν αλλού. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να γίνουν ούτε δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε δικηγόροι, ούτε να πάνε σε ανώτερα ε, εκπαιδευτικά κλιμάκια. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε στη διάθεσή τους ε, για 16χρονους 18 18χρονους και εκπαίδευση ε, τεχνική σε διάφορα επαγγελματικά. Χρειαζόμαστε εξίσου πολύ και μαραγκούς ε, και υδραυλικούς. Και επίση υπάρχει ε, ανάγκη κατάρτιση δασκάλων για να μπορούν να γνωρίσουν τα ταλέντα αυτά του ανθρώπου, για να του καθοδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση. Και ίσω να του βοηθήσει κάποιο να γνωρίσουν άτομα που ίσω εν δυνάμει θα μπορούσαν να καταλέψουν νωρί το σχολείο και να του κατευθύνουν κατάλληλα αλλά βέβαια αυτό είναι θέμα εθνικών, εθνικής αρμοδιότητας των κρατών μελών των Αλλάβων, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε εδώ συζήτηση για να τονίσουμε τα σημεία αυτά, για να προτείνουμε τι θα πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κυρία Χάνιβολ. Δεν ε, μιλάμε για ειδικά ταλέντα και ο Άλμπερτ Άινστάιν δεν ήταν ε, καλός μαθητής αλλά ήταν μεγαλοφυής κι άλλοι μπορεί ε, βέβαια να είναι σε παρόμοια κατηγορία, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι κοινωνικές δυσκολίες και η έλλειψη της ολοκλήρωσης, η ενσωμάτωσης. Είπατε πολλά και σημαντικά, όπως ποιες δυνατότητες δεύτερης ευκαιρίας υπάρχουν πως προβλέπεται συνεργασία μέσα από δίκτυα που έχουν επαφή με αυτούς τους νέους κυρίως, ε, νεαρά αγόρια είναι. Ε, ποιος θα είναι ο ειδικό ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι εμπειρίες υπάρχουν από τα κράτη-μέλη, τι μπορούμε να μάθουμε από όλες αυτές. Στη Γερμανία, στη Βρέμη μας ενδιαφέρουν όλα αυτά αφού είμαστε και υπεύθυνοι εμείς για πολιτική, για τον πολιτισμό, υπάρχει ένα πρόγραμμα για νέους που δεν πηγαίνουν πια στο σχολείο και με καλλιτεχνικά μέσα τους δίνουν μια δυνατότητα έκφρασης για να δουλέψουν αργότερα, να μπουν πάλι σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μετά από έκθεση των έργων τους που θα τα επισκεφθεί το κοινό ε, οι βέλτιστες πρακτικές είναι πολύ σημαντικές για όλη την Ευρώπη. Καλό είναι να μάθουμε τι γίνεται σε άλλους, μην επανεφευρίσκουμε κάθε φορά τον τροχό. Ευχαριστώ. Σομ Κέλλη. Ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστούμε τη Μέρη για την πολύ καλή δουλειά του στο πεδίο. Υποθέτω ότι από ευρωπαϊκή σκοπιά αυτό βρίσκεται στον πυρήνα, αν θέλετε, των αρχών και του τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιτευχθεί ισότητα σε όλα τα κράτη-μέλη στο θέμα και ιδιαίτερα προσπάθεια να βοηθήσει τα άτομα να τύχουν κάποιε εκπαίδευση, γιατί γίνεται όλο και πιο σημαντικό το θέμα τη παιδεία, να υπάρχει παιδεία ιδιαίτερα στην ε, εποχή που ζούμε και ιδιαίτερα με την αναζήτηση νέων δεξιοτήτων και νέων θέσεων απασχόλησης γιατί εάν δεν έχουν νέε δεξιότητε, όλο και λιγότερε πιθανότητε θα έχουν να βρουν ε, απασχόληση τα νέα άτομα. Και βέβαια, όσοι εγκαταλείπουν όλοι στο σχολείο έχουν όλο και περισσότερε πιθανότητε να εμπλακούν σε αντικοινωνικέ δραστηριότητε και συμπεριφορέ. Αυτό είναι στόχο κλειδί λοιπόν το 2020. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε πολύ πιο σκληρά γι' αυτό, γιατί τα ωφέλη θα είναι τεράστια σχετικά. Μια πτυχή που θα ήθελα να τονίσω είναι κάτι που φαίνεται να επηρεάζει πολύ περισσότερο τα αγόρια από τα κορίτσια. Τα αγόρια καταλήγουν νωρίτερα το σχολείο από τα κορίτσια και νωρίτερα και με μεγαλύτερη συχνότητα. Ένα από τα σημεία κλειδιά λοιπόν είναι η επένδυση που γίνεται για τα παιδιά νεαρής ηλικία, Όσο νωρίτερα, όσο επενδύουμε σε νεότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερε οι αποδόσει. Αυτό είναι κάτι πάγιο, δεδομένο. Πρέπει να δούμε την επένδυση, εξίσου σημαντική επένδυση στην προσχωρική ηλικία και στο, και δημοτικό. Και αυτό μπορεί να φέρει άρδιν διαφορετική προσέγγιση στην προσέγγιση των παιδιών. Και ίσω θα πρέπει να υπάρχει οικονομική δέσμευση των κρατών μελών. Γιατί αυτοί που εμπλέκονται ε, σημαντικά στην προσχολική παιδεία, κατά κύριο λόγο είναι εις των γονέων. Πρέπει να, αυτοί που ασχολούνται με τα παιδιά, αν θέλετε, σε προσχολική ηλικία είναι περισσότερο ανήλικες, ανήλικα μέλη της οικογένειας, ενώ οι γονείς λείπουν για δουλειά. Εάν ψάξουμε λοιπόν να βελτιώσουμε τα προσόντα των ανθρώπων που ασχολούνται αυτή τη ηλικία και βάζοντα την έμφαση εξίσου σε άνδρες και γυναίκες. Μέχρι στιγμή η έμφαση που δίνεται σε αυτό το επίπεδο ήταν σε γυναίκες, αν θέλετε, νηπιαγωγούς εμπλεκόμενες στην προσχολική ηλικία. Σε πολλές χώρες υπάρχουν πολύ πετυχημένα προγράμματα αλλαγής του υποδείγματος, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, όπου στη Δανία έχουν ε, ε, εγκρίνει και έχουν φτάσει το 25% ανδρών να ασχολούνται με προσχολική ηλικία. Αυτό είναι πολύ καλό για την αλλαγή των μοντέλων και να υπάρχει ισορροπία. Και βέβαια με σωστή εκπαίδευση και απολαβέ μπορεί να επιτευχθεί, γιατί αν υπάρχει σωστή κατάρτιση, προφανέστατα πολλά από αυτά που θέλουμε να πετύχουμε δεν πρόκειται να επιτευχθούν. Δεύτερον, σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη φάση, τα παιδιά κάνουν πράγματα φυσικό το τρόπο. Δεν ασκείται πίεση ή στρες πάνω τους. Αν δημιουργηθεί λοιπόν το σωστό κλίμα στην νεότερη δυνατή ηλικία, θα μπορεί να μεταφερθεί αυτό και στο ε, πιο τυποποιημένη θέλετε, και επίσημη εκπαίδευση, ε, δημοτικό και μετά. Και αυτό θα βοηθήσει να δημιουργήσει μια θετική εικόνα. Και τα ωφέλεια στη συνέχεια θα είναι τεράστια από πλευράς ε, κοινωνίας. Χωρίς να μπω λοιπόν σε λεπτομέρειες, γιατί θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε με τις τροπολογίες και στην όλη διαδικασία που θα ακολουθήσει, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το φαινόμενο αυτό, πολύ σημαντικό στόχος που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν καταφέρουμε λοιπόν όντως να μειώσουμε μόνο στο 10% το ποσοστό αυτών που εγκαταλείπουν νωρίτερα το σχολείο, θα διευκολύνουμε πολύ την ζωή όλων των Ευρωπαίων πολιτών και εν κατακλείδη να βελτιώσουμε ευρύτερα την ευρωπαϊκή οικονομία. Ελπίζω λοιπόν να μπορούμε να σηματοδοτήσουμε, να φέρουμε, σημαντική πρόοδο με την εμπλοκή μας αυτό. Ευχαριστούμε. Λόταρ Μπίσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο, μεγάλη προσοχή την έκθεσή σας, την παρουσίαση. Συμφωνώ με πολλά. Ε, θέλω να αναφερθώ στη δεύτερη ευκαιρία. Είναι σωστό να υπογραμμίζουμε τη δεύτερη εμπειρία. Αυτό ε, στηρίζεται στην εμπειρία. Και παλιότερα και ακόμα τώρα ε, ασχολήθηκα με τους καλλιτέχνες που μετά την πρώτη, δεύτερη, στην τρίτη προσπάθεια γίνονται επιτυχημένοι καλλιτέχνες. Υπάρχουν πολλά που τεκμηριώνουν ότι μετά από πολλές προσπάθειες ε, πέτυχαν και καταξιώθηκαν. Είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την υποδομή για τη δεύτερη και την τρίτη θα έλεγα εγώ ευκαιρία. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα με τις ε, υπεύθυνε επιτροπές και τη σύνθεσή τους που μπορεί να είναι δημοκρατική αλλά μπορεί παράλληλα να παραβλέπει και κάποια μεγάλα ταλέντα. Στο Ποτστάμ έπρεπε πολλές φορές να ε, κάνουμε νέα σύνθεση στις επιτροπής και ξαφνικά προέκυψαν καινούργια εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ε, νέοι καλλιτέχνες, σκηνοθέτες κλπ όλα τα κοινωνικά αίτια που λέτε είναι σωστά να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τη δεύτερη ευκαιρία και την τρίτη. Γιατί υπάρχουν ταλέντα που αναδεικνύονται σε διαφορετική ηλικία κάθε φορά. Παίζουν ρόλο και το φύλλο εδώ. Πολλές φορές η οριμότητα έρχεται νωρίτερα στις κοπέλες από ό,τι στα γόρια ή ε, μπορεί άλλα να παίζουν ρόλο για την ηλικία που θα ε, αποκαλυφθεί ένα ταλέντο. Γι' αυτό να δίδεται και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Μέσα από την προοπτική κάποιου που τα έζησε αυτά και από το σχολείο, πράγματι είναι καλό να υπάρχουν ευκαιρίες. Και τέταρτη ακόμα, να υπάρχουν άνθρωποι με ευρύς ορίζοντες και όχι με παροπίδες ε, δεν θέλουμε μειοπική δηλαδή αξιολόγηση. Και ο κύριος Τάπιο Σαράλα από την Κομισιόν εάν επιθυμεί. Ε, είναι από τον τομέα της εκπαίδευσης, της σχολικής εκπαίδευσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι η μείωση της προώρης εγκατάλειψης του σχολείου είναι ένας από τους στόχους της στρατηγικής του 2020 και έχει επιπτώσεις και σε άλλους στόχους που αφορούν την απασχόληση και τη μείωση της ανέχειας στην Ευρώπη. Όπως είπαν πολλοί ομιλητές, η πρόορη κατάληψη του σχολείου έχει τρομερές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων, στις οικογένειές τους και στα παιδιά τους. Γιατί μειώνει τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι το ευρωπαϊκό κριτήριο της μείωσης ε, του αριθμού των προώρως εγκαταλειπώντων σε 10% μέχρι το 2020 είναι κάτι που όπως ξέρετε επαναλαμβάνεται γιατί είχε ξαναϋποθεί και δεν επετεύχθη ο στόχος το 2010. Επίσης το 17,4% αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο το έχουν εγκαταλείψει από το δημοτικό ήδη. Για να σας δείξω λιγάκι ποια είναι η επίπτωση αυτού του φαινομένου, θα έλεγα ότι αν μπορούσαμε να μειώσουμε κατά 1% τον αριθμό των προώρως εγκαταλειπώντων, θα δημιουργούνταν έτσι 500.000 περισσότεροι ε, ειδικευμένοι εργαζόμενοι στο δυναμικό μας. Πρέπει καταρχήν να καταλάβουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Γι' αυτό προτείναμε ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτικής με αντισταθμιστικά μέτρα και παρέμβαση, αλλά επίσης τονίζουμε ότι χρειάζομαστε πολύ ακριβέστερα στοιχεία και δεδομένα σε πανενωσιακό επίπεδο για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει μάλιστα να πω ότι υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα βελτίστων πρακτικών, αλλά η κύρια πρόκληση είναι πώς θα δημιουργήσουμε συνεπή και συνολική πολιτική, διότι η πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου είναι, όπως είπατε και εσείς, πολύπλοκο φαινόμενο και γι' αυτό χρειάζεται πολύπλοκη αντιμετώπιση. Πολύ συνεργασία, κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερομένων και παραγόντων. Άρα, δεχόμαστε την πρωτοβουλία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή τη γνωμοδότηση, και φυσικά προσμένουμε στην, ε, μπορείτε να υπολογίζετε στη βοήθειά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Σε σχέση με αυτό το θέμα της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου, μετά την τελευταία συζήτηση, η κυρία Βασιλείου έκανε μια συνάντευξη τύπου μετά την ανακοίνωση και ζήτησαν δημοσιογράφη να αποφανθώ. Διαπιστώθηκε ότι δεν είναι αρμόδια. Θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε την ανακοίνωση, την όλη διαδικασία, την ανασχόληση του Κοινοβουλίου, τη γνωμοδότηση. Δηλαδή όλα αυτά δημιούργησαν μια ε, ε, αφύπνιση για το πρόβλημα οι συνάδελφοι Μπίσκι, Τρούπελ και άλλοι είπαν ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα εδώ και δεν είναι εύκολο να γίνει η ανταλλαγή τους. Χρειάζεται μια πλατφόρμα οργανωμένη. Δεν θα πάμε στον μπαρ να τα λέμε αυτά. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνόδους των Υπουργών έχει μια πλατφόρμα. Αλλά μέχρι να μπουν όλα αυτά στα κεφάλια των δημοσιογράφων περνάει χρόνος. Γιατί μ' άκουσα να μιλάω και είπαν κυρία Πακ, τι είναι αυτά, δεν υπάρχει κάποια, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Πολλά και πάρα πολλά είπα εγώ, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη αν δεν ε, ξέρετε ας πούμε το θαυμάσιο παράδειγμα της Βρέμης ε, που καλό θα ήταν το παραθέσω και εγώ ή άλλα παραδείγματα αν δεν τα ξέρετε αυτά σας λείπει μια εμπειρία που θα σας βοηθήσει και σας να δραστηριοποιηθείτε πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που η Κομισιόν κάνει σε αυτούς τους τομείς πράγματα τα οποία δεν ε, είναι επιβεβλημένα να τα κάνει με βάση τη συνθήκη που όμως δημιουργούν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τις βέλτιστες πρακτικές. Καμιά φορά οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να καταλάβουν την αξία του έργου αυτού της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και σε αυτό το τομέα και σε άλλους τομείς, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού κλπ. Αυτά τα καταληκτικά είχα να πω. Η κυρία Χάνιμπολ θέλετε να πείτε κάτι. Ναι. Να ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά τους και για αυτά που μόλις είπατε που συνοψίζουν την προσέγγιση που πρέπει να έχουμε. Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία στο θέμα αυτό, γιατί για να είμαι, αν θέλετε, κατηγορηματική και ομή, τα στοιχεία τα οποία βλέπω με πρόορη εγκατάλειψη σχολείου είναι πραγματικά σοκαριστικά. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Το θέμα είναι έντονο κοινωνικό, αφορά μεν στα άτομα, αλλά είναι και ένα πολύ ευρύτερο οικονομικό ζήτημα. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά και σημείωσα όλα τα σχόλια που έκαναν οι πάντες στην έκθεση αυτή. Πρέπει να βγούμε, να παλέψουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ευχαριστούμε. 15 Ιουνίου θα συζητηθεί το προσχέδιο της έκθεσης και θα ψηφίσουμε στις 14 Ιουλίου. Ερχόμενοι τώρα στο σημείο 15, την απόφαση των συντονιστών. Συζήτησα σήμερα το πρωί, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, ελπίζω να εγκρίνεται. Αυτά που ζητήθηκαν. 16 τα διάφορα. Τίποτα. 17. Επόμενη ημερομηνία 25 και 26 Μαΐου. Και ευχαριστώ τους Δερμηνείς που έχουν πλέον ελεύθερη χρόνο. Χάνει την απουσία της κυρίας Βασιλείου και τον Πρόεδρο.